Παρακαλώ να ζητήσω από τους συναδέλφους να καθίσουν. Καθίστε παρακαλώ να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Να καλωσορίσω την κυρία Ντανιέλ Νουή, πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Εποπτικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε εδώ και αρκετό καιρό. Τα είπαμε στις 26 Μαρτίου επί τη ευκαιρία της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου. Σήμερα είναι η πρώτη τακτική δημόσια κρόση που έχει προβλεφθεί για το 2018 στο πλαίσιο της Διοργανικής Συμφωνίας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα κρίσιμα ζωτικής σημασίας που θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα. Ξέρουμε ότι στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις θα ασχοληθείτε με αυτά τα θέματα. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Single Rule Book, γιατί αργότερα ελπίζουμε στις 6.30 ότι θα ψηφίσουμε για τη δέσμη μέτρων για τον τραπεζικό τομέα, το οποίο αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. και για το Single Rule Book, αλλά και για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων που αποτελούν και το πλαίσιο εργασίας μας. Έτσι κάνουμε ένα βήμα παραπέρα για τη μείωση του κινδύνου κάτι το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα και χαιρόμαστε κυρία Νουή που είστε εδώ μαζί σας. Έχετε ευθύ αμέσω το λόγο για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως πάντοτε, είναι μεγάλη χαρά για μένα που έχω την ευκαιρία να σας επευθύνω το λόγο σήμερα, να ακούσω τις ερωτήσεις σας, τις ανησυχίες σας και να συζητήσω το ρόλο μας ως ε, Εποπτικό Συμβούλιο τη ΕΚΟΥΤΟΥ. Θα ε, ασχοληθώ με την Targeted Review για... ε, ε interim models για τους κινδύνους κυβερνοαπειλές, για το Brexit και για τους βασικούς νομοθετικούς φακέλους. Θα σας ενημερώσω και για την πρόοδο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πολύ σημαντικές είναι οι πρόοδοι που έχουμε επιτύχει για την αναθεώρηση αυτών των μοντέλων. Έχουμε ερευνητικά σχέδια και για το, την περίοδο 2017-2019 να αξιολογήσουμε κατά τα πόσο είναι αρκετά τα internal models, τα εσωτερικά πρότυπα που υιοθετούν οι τράπεζες της κατηγορίες τύπου 1. Το TRIM λοιπόν έχει ήδη φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Έχουμε κοινή κατανόηση μεταξύ των τραπεζών, των προαπαιτούμενων που είναι εφαρμοστέα από την νομοθεσία για τα εσωτερικά μοντέλα που έχουν στην ζώνη του ευρώ και όλα αυτά φαίνονται στον λεπτομερή οδηγό που έχουμε στην ιστοσελίδα μας. Χάρη στην αναρμονισμένη μεθοδολογία και τα εργαλεία τα σχετικά με το τρίμ έχουμε οριζόντια ανάλυση συγκρίσεις μεταξύ ομολόγων και έγκαιρα βλέπουμε πού είναι τα εμπόδια και δεν μπορεί μια τράπεζα να συμμορφωθεί με την νομοθεσία όποτε αυτό συμβαίνει και μπορούμε έτσι να λάβουμε και αποφάσεις κατάλληλες και να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες εφαρμόζουν την νομοθεσία στα εσωτερικά τους μοντέλα, τα internal models. Είναι προφανές ότι ενημερώνουμε τις τράπεζες για το project αυτό συνεχώς και σημειώνουμε σημαντική πρόοδο και στα stress test των τραπεζών τα φετινά. Θέλουμε να αποπτεύουμε τις τράπεζες και να έχουμε ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο να συγκρίνουμε την ανθεκτικότητα και την αντοχή των τραπεζών στα διάφορα σοκ της οικονομίας, κατά πόσο μπορούν τα σοκ αυτά να θέσουν σε κίνδυνο την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Θέλουμε για τον κίνδυνο φερεκιότητας των τραπεζών να κάνουμε σωστά τεστ για ε, τα χειρότερα δυνατά σενάρια, ε, conduct risk, operational risk, market risk, μεταξύ άλλων αλλά θέλουμε να δούμε και πώς αυτό επηρεάζει τα έσοδα από τις προμήθειες. Τα stress test μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες που συλλέγουμε, τα χρησιμοποιούμε για να έχουμε αξιολόγηση της κατάστασης της κάθε τράπεζας. Μιλούμε για 33 τράπεζες στη ζώνη του ευρώ και για αυτές τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στις 2 Νοεμβρίου φέτος. Για τις ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα stress test η άσκηση υιοθέτησε την ίδια μεθοδολογία με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έγινε με επιταχυμένο χρονοδιάγραμμα πριν από, την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής ε, ε, προσαρμογής για την Ελλάδα. Τα stress test για την Ελλάδα έδειξαν ότι έχουμε νέα ποσοστιαίες μονάδες στην, ε, ε, σε σχέση με τη κεφαλιακή επάρκεια 15,1 δις στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Είχαμε παραμέτρους για τον πιστοτικό κίνδυνο και το καθαρό εισόδημα από τόκους και επιτόκια. Για τους κυβερνοκινδύνους και κυβερνοαπολές καλωσορίζουμε τις διεθνείς προσπάθειες που έχουν γίνει να υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και γνώση. Όλο και περισσότερο ψηφιοποιείται η τραπεζική. Άρα εξελίσσεται και οι κυβερνοαπειλές που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Έχουμε αλληλεξάρτηση με εξωτερικούς παρόχους τεχνολογίας της επικοινωνίας και πληροφοριών. Έχουμε όλο και πιο εξελιγμένους και περίπλοκους κυβερνοκινδύνους. Και μας ενδιαφέρει πολύ αυτός ο τομέας. Έχουμε εστιάσει τις προσπάθειες μας σε αυτό το επίπεδο και θέλουμε οι τράπεζες να ιεραρχήσουν τις απειλές και να έχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας εσωτερικό και μεγάλη επαγρύπνηση. Θέλουμε να ε, υπάρχει γρήγορη αντίδραση στις απειλές που αναδύονται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι τράπεζες είναι ασφαλείς και α, έχουν πλήρη ανοσία. Θέλουμε να συνειδητοποιήσουν ότι πάντοτε πρέπει να αντιμετωπίζουν κυβερνοαπειλές και να είναι πάντοτε σε εγρήγορση και σε κατάσταση ετοιμότητας. Τώρα, οι περισσότερες τράπεζες που είναι υπό την εποπτεία της ΕΚΟΤΟΥ ε, προοδεύουν και προσαρμόζονται στο περιβάλλον μετά το Brexit. Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία να τροποποιήσουν την παρουσία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και να έχουν την απαραίτητη αδειοδότηση από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από την αναθεώρηση των σχεδίων τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για τις τράπεζες που μετεγκαθίστανται στη ζώνη του ευρώ δεν έχουν ακόμα υποβάλει αίτημα για αδειοδότηση και τελειώνει ο χρόνος τους. Τους ζητούμε να μας υποβάλουν αιτήσει πριν από το τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2018. Οι τράπεζες που δεν έχουν υποβάλει πλήρη αιτήματα και πλήρης φακέλους πρέπει να γνωρίζουν ότι ίσως δεν πάρουν έγκυρη διαδότηση για να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την τραπεζική τους δραστηριότητα μετά το Brexit. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τα σχέδιά τους και τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα εφαρμόζουν γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ε, τράπεζες που τελικά είναι άδεια και δεν μπορούν να διεξάγουν σωστή τραπεζική δραστηριότητα. Για την Τραπεζική Ένωση θεωρούμε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση κινδύνου και άρα μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο και πρόγραμμα κοινή εγγύησης καταθέσεων και να έχουμε common backstop ε, για το ενιαίο ταμείο για την εξυγίαση και διάσωση των τραπεζών μπορεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση εγκαίρως και καλωσορίζουμε το γεγονός ότι το Συμβούλιο θέτησε τη γενικότερη προσέγγιση του το Μάιο και περιμένω να εγκριθούν οι εκθέσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει γρήγορα ο τριμερής διάλογος για να μπορέσει να ευθετηθεί αυτή η δέσμη μέτρων αρκετά πριν τις επόμενες ευρωεκλογέ. Το Μάιο του 19 για τις, ε, ε, τα ελάχιστα ε, προαπαιτούμενα για το MRL. Χαίρομαι διότι διαγράφηκε το guidance για το MREL και επεκτάθηκαν οι περίοδοι συμμόρφωσης. Η αναθεώρηση του MREL θα ετονίσει την μεταστροφή από το bail-out προς το bail-in τη διάσωση με ίδια κεφάλαια και ίδιους πόρους. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να μειωθούν εσωτερικά τα MRL και αυτό θα είναι ένα τρόπος να λειτουργήσουν και οι θυγατρικές ε, τράπεζες. Υπό τον όρο ότι υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές ε, δικλίδες έτσι ώστε να υπάρχει στήριξη από τη μητρική εταιρεία στην θηγατρική. Θα έχουμε χαμηλότερα κατόφλια και καλύτερη κατανομή των πόρων εντός του ίδιου τραπεζικού ομίλου. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, στην κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος επίσης. Τώρα, για να λειτουργήσει αυτό, πρέπει να έχουμε απρόσκοπτη κεφαλιακή ροή σε δύσκολες περιπτώσεις. Και αυτό θα αντικατοπτρίζει το ότι μιλούμε για μία και μόνη ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση. Γνωρίζω ότι κάποιες προτάσεις εξετάζονται για απόκληση από τα πρότυπα της Βασιλείας προτινόμενες αλλαγές στη μεθοδολογία της Βασιλείας για να υπολογιστεί ο λόγος του μόχλευσης. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να διασφαλίσουμε ότι γενικά οι τράπεζες συμμορφούνται με την νομοθεσία και υπάρχουν ίσες συνθήκες και προϋποθέσεις για όλους. Είναι σημαντικό οι υποπτικές αρχές να μπορούν να αποφασίσουν για τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η κεφαλαιακή σύνθεση η σύνθεση του κεφαλαίου, των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση καλωσορίζω το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Να μειώσουμε τις εθνικές επιλογές ε, της διακριτικής ευχέρειας και αντιμετώπισης. Και επίσης Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση των εθνικών πλαισίων για να κηρυχθεί μια τράπεζα φερέγγια ή αφερέγγια. Έτσι θα έχουμε παιχνίδι επίσης όρης και θα είναι πιο αποτελεσματική η δουλειά της εκάστοτε εποπτικής αρχής. Πάρα πολλέ και περίπλοκε επιχειρήσει αυτή τη στιγμή σχεδιάζουν να επενδύσουν και να εγκατασταθούν στη ζώνη του ευρώ μετά το Brexit ω επενδυτικέ εταιρείε και επιχειρήσει. Καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να έχουμε ένα στεναρό πλαίσιο, να μην έχουμε αυξημένο κίνδυνο και να μην έχουμε και κίνδυνο spillover. Να, να υπόκεινται αυτές οι επενδυτικές επιχειρήσεις στο ίδιο νομικό πλαίσιο όπως τα πιστατικά ιδρύματα και τα χρηματοπιστατικά ιδρύματα. Αυτό ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι δεν έχουμε κατακαιρματισμό της νομοθεσίας και ε, παράγοντες και εταιρείε που δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στον ίδιο τομέα να υπόκεινται η κάθε μία σε, σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Τώρα, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια... Που βεβαίω είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό για το ευρωπαϊκό σύστημα θέμα. Έχουμε σημαντική πρόοδο χάρη στην ευρύτατη δουλειά που έχουν κάνει οι εποπτικέ αρχές. 60% και άνω του συνολικού ποσού των μη εξυπηρετημένων δανείων τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει εξασφαλιστεί χάρη στο, στις του 2017. Έχουμε τελικά... Έχουμε δημοσιοποιήσει την τελική μας έκθεση το Μάρτιο για τη διαμόρφωση των ε, συνθήκων στα νέα με εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχουμε τους οδηγούς προς τις τράπεζες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και δεδομένου ότι είναι πιο θετικές οικονομικές εξελίξεις. Οι νομοθετικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις ε, ρυθμιστικές αρχές και την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων είναι πολύ σημαντικές, υπάρχει συνεργασία στο θέμα της εξυπηρέτησης, της αντιμετώπισης μάλλον του αποθέματος με εξυπηρετουμένων δανείων συνεχίζει τη δουλειά. Βεβαίως θέλουμε να συστήσουμε σε στις λεπτομέρειες αργότερα και καλώς ορίζω βέβαια τις ερωτήσεις σας για τα θέματα αυτά. Κύριε Ντελάνγκη, έχει το λόγο. Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις θέματα, αν θέλετε. Καταρχάς, για την υπόθεση ABLV. Και ξέρω ότι δεν είναι καθαρά ζήτημα δικών σας αρμοδιοτήτων, αλλά οπωσδήποτε η νομιμοποίηση παρανομών εσόδων, το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα σοβαρό θέμα. Έχετε δηλαδή και ρωτώ κάποιο τρόπο να παρακολουθήσετε αυτές τις εξελίξεις, να σας επισημένονται κάποιες υποθέσεις ίσως ταχύτερα και τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο για να αλλάξει αυτό. Ή, επί παραδείγματι, τι είδου δείκτε πρέπει να παρακολουθεί κανεί. Βλέπετε να υπάρχουν περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με μεγαλύτερο αριθμό πελατών που είναι μη κάτοικοι ή πάντως όχι διαμένονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην είναι βέβαια θέματα του ίδιου, αλλά όταν έχουμε μεγάλο αριθμό ε, καταθέσεων ή μεγάλη βάση καταθέσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασφαλώς ε, ο κίνδυνος πρέπει κάπως να επισημαίνεται στο ίδις. Και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Φαντάζομαι θα περιμένατε την ερώτησή μου, μια και εσείς το φέρατε το θέμα ε, πιο, για πιο μετά, δηλαδή το αναβάλατε για μια επόμενη συνεδρίαση. Ε, όταν έχουμε λοιπόν ένα εφιστάμενο δάνειο, το οποίο από μια στιγμή και μετά πάβει να εξυπηρετείται, για να ξεκαθαρίσουμε τουλάχιστον αυτό, αν δεν θέλετε να δούμε τις λεπτομέρειες τώρα, μπορείτε παράλληλα να εξετάσετε πόσο στεναρός είναι ο τραπεζικός τομέας στον τομέα αυτών Πώς μπορούμε να κοιτάξουμε τα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα, από ένα σημείο και μετά υφιστάμενα που μετατρέπονται σε μη εξυπηρετούμενα. Και οπωσδήποτε αυτό ενδιαφέρει την Επιτροπή. Αν έχετε έστω μια μικρή ιδέα για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, με ενδιαφέρει πολύ να το ακούσω. Αλλά η πρώτη μου ερώτηση ήταν και η πιο σημαντική. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Σε σχέση με την ε, κατάσταση σχετική με την ε, ABLV. και τη δυνατότητα για πιο έγκαιρη παρέμβαση η αντίδραση. Οπωσδήποτε η νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομοποίησης παρανόμου χρήματος θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον δεν είναι παντού ξεκάθαρο, το τι μπορούν να κάνουν οι δημόσιες αρχές που επιλαμβάνονται της καταπολέμησης της νομοποίησης παρανομών εσόδων, κυρίως όσον αφορά την κοινοποίηση σε στοιχεία, στοιχεία που θα ήταν και το μέσο για να μπορούσαμε να αντιδράσουμε ταχύτερα. Αυτή η δυνατότητα, δηλαδή ανταλλαγής απόρριτων στοιχείων, φαντάζομαι ε, θα καλυφθεί οπωσδήποτε με την νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομοποίησης παρανομών εσόδων. Εγώ προσωπικώς θα προτιμούσα να είχαμε μορφή κανονισμού και όχι οδηγίας, γιατί η οδηγία πρέπει να περάσει στην εθνική νομοθεσία και μεταφέρεται με πολλούς και διάφορους τρόπους και σε εκ τούτου δεν είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τους στόχους της. Μετά, έχετε ε, ερώτηση, μου λέτε, εάν, ε, ε, με ρωτάτε αν έχουμε υπόψη κάποιες τράπεζες που έχουν μεγάλο ποσοστό καταθέσεων που δεν εδράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως έχουμε ει βάθο γνώση των δραστηριοτήτων των τραπεζών και βεβαίως ω προ τη συγκεκριμένη σα ερώτηση έχουμε πολλή δουλειά κάνει με τα Υπουργεία Οικονομικών, με τις εποπτικές αρχές, συνεργασία με τις λοιπές εθνικές αρχές, τις αρμόδιες για την καταπολέμηση τη νομιμοποίησης παράνομου χρήματος, ώστε να μειώνεται ο αριθμός αυτή η βάση καταθετών που δεν έχουν διαμονή, ε, μάλλον κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μειώνεται ουσιαστικά του λεχθέντο. λεχθέντος. Εμείς αρμόδιοι για τη σχετική οδηγία, για την καταπολέμηση δηλαδή παρανόμου χρήματος, δεν έχουμε. Και άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σαν πανέμβαση είναι να συνεργαστούμε με την Εθνική Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμου χρήματος. Αλλά δεν έχουμε πάντα τα στοιχεία, δεν μας ε, μεταδίδονται, δεν... Ε, καλύπτεται πάντα αυτό το θέμα της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών για τα απόρριτα δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε, όταν εξουσία άλλοι δεν έχουμε παρά μόνο την πειθό, προσπαθούμε να πείθουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και για τις αρχές αυτές να μας ενημερώνουν και ότι μπορούν να γίνονται και επιτόπιες έρευνες στις τράπεζες που κρίνονται υποπτέ, Όχι ότι οι ίδιες νομιμοποιούν ε, παράνομο χρήμα, αλλά ότι αυτές τις επισκέψεις ε, θέλουμε να τις κάνουμε για να βεβαιωνόμαστε ότι δεν χρησιμοποιούνται οι τράπεζες από κάποιους που θέλουν να ξεπλύνουν χρήμα. Και άρα προσπαθούμε να πείσουμε ότι είναι και για τις ίδιες καλό αυτό, αυτός ο έλεγχος που γίνεται. Πάντως στην Ευρώπη η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από τις σε άλλα μέρη του κόσμου. Για το απόθεμα τώρα μη εξυπηρετουμένων δανείων. Καταρχάς επιμένω στη δουλειά που έχουμε κάνει. Έχει ήδη αρχίσει να φέρνει καρπούς. Ξεκινήσαμε το 2014 με ένα με ένα 3 εκατομμύριο ε, σε έκθεση και φτάσαμε στα 670 δισεκατομμύρια το 16 ε, με 17. Αλλά ε, όσο και αν είναι πολλά τα 670 δισεκατομμύρια, οπωσδήποτε η μείωση από το 1 τρισεκατομμύριο είναι πολύ σημαντική. Από το 7% έχουμε πέσει στο 4,9%. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν ποσοστό. Βέβαια, ανάλογα με την τράπεζα ή το τραπεζικό σύστημα, γιατί εκεί περιπλέκονται τα πράγματα. Μετά συμφωνώ ότι πρέπει να ε, ε, την χάνουν ίδια αντιμετώπιση όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρέπει ο ίδιος κίνδυνο να έχει την ίδια αντιμετώπιση πάντα. Είτε πρόκειται για καινούργιο δάνειο με εξυπηρετούμενο, είτε πρόκειται για δάνειο που εξυπηρετούνταν, αλλά άρχισε να μην εξυπηρετεί από ένα σημείο και μετά. Ο κίνδυνο, όπω λέω, είναι ο ίδιο και πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση, αλλά ε, πρέπει να είμαστε και Εάν το πρόβλημα έχει περιορισμένε διαστάσει, ίσω χρειάζεται λιγότερη ένταση προσπάθειας από ότι ένα πρόβλημα που έχει μεγαλύτερε διαστάσει. Πάντως προσπαθούμε και με την επικοινωνιακή μας πολιτική και ανακοίνωση και τα λοιπά που θα κάνουμε να εξηγούμε πού έχουμε φτάσει, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. έτσι ώστε να καταστεί και για τις τράπεζες πιο ξεκάθαρη κατάσταση. Βήμα το βήμα, αλλά έχουμε και τις ασφαλιστικές δικλίδες. ώστε να εξασφαλίσετε ότι πράγματι αυτή η δράση που αναλαμβάνουμε είναι και ρεαλιστική. Υπέρ Μπέρα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Θα θέλαμε να επανέλθουμε ε, σε ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πολύ συχνά από τη στιγμή που ε, οι ε, Αμερικάνοι αποκάλυψαν τον προβληματισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπάθησε να δουλέψει για τη βελτίωση του BRD. Η Κεντρική ιδέα είναι ότι μάλλον θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στι εθνικέ αρχές οι οποίες ε, ε, ε, καταπολεμούν, έχουν αναλάβει την καταπολέμηση κατά του ξεπλήματος χρήματος να αντιμετωπίσει το θέμα. Θα πρέπει βέβαια να δούμε σε ποιο ακριβώς επίπεδο βρίσκεται η καταπολέμηση της νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων στις διάφορες χώρε. και βεβαίω αυτό ξεπερνά κατά πολύ την εντολή αλλά ε, βεβαίως εσείς για να μπορέσετε να υλοποιήσετε τις λεπτομέρειες ε, και τα επιμέρους στοιχεία της εντολής σας πρέπει να ξέρετε και πώς έχει το κλίμα γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να ξέρετε τι κάνει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Η ερώτησή μου αφορά στην ουσία την, την διακυβέρνηση των δομών, των τραπεζικών δομών, ε, γιατί ούτε ε, το επίπεδο ένα της δομοθεσίας ούτε όμως ε, και οι συνθήκες αναφέρουν λεπτομερώς την διάρθρωση της διακυβέρνησης, παρά μόνο εάν πρόκειται για κάποιες τοξικές δομές και ε, ε, σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η διαφοροποίηση από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και κάποιες δομές οι οποίες δεν είναι καθόλου συμβατές με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά δουλεύοντας πάνω σε θέματα με το SSM και το OPA βλέπουμε ότι ακολουθούμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες με την αιτιολογία ότι σε ορισμένες συνεργατικές διαδικασίες ε, μπορεί να υπήρξαν προβλήματα, ε, μας οδηγεί σε καταστάσεις οι οποίες είναι περίεργες. Δηλαδή για μεγάλες συνεργατικές ε, ε, δομές ε, ή άλλου είδους αμοιβαιότητας δίνεται η αλληλασφάλισης, δίνεται η δυνατότητα να απλουστεύσουν κάποια πράγματα. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι γενικά θα έπρεπε να απλουστευτεί η κατάσταση σε ένα ενιαίο μοντέλο, έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα να εφαρμοστεί. Ο στόχος όμως ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ή ο στόχος της δικιάς σας εντολής είναι εν τέλει αυτός. Ε, Θα σας απαντήσω στα αγγλικά έτσι ώστε να καταλάβουν ε, καλύτερα οι περισσότεροι. Πρώτον, όσον αφορά το ξέπλυμα και την, την νομοθεσία σχετικά με αυτή την νομοποίηση παρανόμων εσόδων είναι γεγονός ότι ας πούμε η Λετωνία που είναι μια μικρή χώρα με μικρή εποπτική αρχή που έχει εξουσίες που αφορούν και το θέμα ε, της ε, νομιμοποίησης ε, παρανόμων εσόδων, έχουν συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού και λόγω της παγκοσμιοποίησης αντιμετωπίζουν και αυτή κίνδυνο παρότι είναι μικρή και μακριά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε στην Ευρώπη. Μια οργάνωση όπως είναι το SSM, όπου υπάρχει ε, μια υπηρεσία που μπορεί να βρίσκεται στις Βρυξέλλες ή στη Γερμανία ή στη Φραγκφούρτη ή κάπου αλλού ε, αλλά και κάποιες ε, άλλες αρχές γύρω, γύρω τριγύρω οι οποίες μέσω της εθνικής πραγματογνωμοσύνης μέσω των διασυνοριακών επιθεωρήσεων μπορούν με πιο επιτυχή τρόπο να ολοκληρώσουν την όλη διαδικασία. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως Χρειάζεται οπωσδήποτε και ισχυρή νομοθεσία ε, οι οδηγίες ε, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία με 50 διαφορετικούς τρόπους ε, δεν είναι το καλύτερο εργαλείο και λυπούμε που θα έχουμε ένα νέο, μια νέα οδηγία και όχι κανονισμό που θα έδινε την δυνατότητα μιας ισχυρής ευρωπαϊκής προοπτικής. Πάντω τα προβλήματα ούτω ή άλλως δεν μπορούν να εξαφανιστούν, τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα βάλουμε ε, κάτω από το χαλί και κατά την ε, δική μου προσωπική άποψη ε, δεν είναι η καλύτερη λύση η επιλογή της οδηγίας. Όσον αφορά τις τραπεζικές δομές, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας πω ότι ε, ακριβώς λόγω προσέκουσης νομοθεσίας ε, και ε, ενός γενικού νομοθετικού πλαισίου μέσω άλλων οδηγιών που προβλέπουν μια ελάχιστη εναρμόνιση αλλά μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά την ε, εφαρμογή ε, ε, ναι θεωρώ ότι δεν είναι η θετική ποικιλομορφία που θα έπρεπε να έχουμε όσον αφορά την ίδια την ε, διακυβέρνηση, δηλαδή τράπεζες ε, σε αντιδιαστολή με, την, ε, με τις υπηρεσίες ή τα ταμεία αλληλασφάλισης, τράπεζες σε αντιδιαστολή με τις συνεργατικές τράπεζες. Κοιτάξτε, εμάς μας αρέσει η διαφοροποίηση, μας αρέσουν διαφόρων μορφών τράπεζες, μεγάλες, μικρές, μεσαίες. εγώ είμαι απολύτως πεπισμένη ε, ότι ο τρόπος με τον οποίο ε, έχουμε εφαρμόσει ε, τις διάφορες νομοθετικές αρχές στα πλαίσια του CCM και από πλευράς του κλάδου, από τις δημόσιες τράπεζες, τις ιδιωτικές τράπεζες, οι τράπεζες αλληλασφάλισης, οι υπηρεσίες αυτές, όλοι, όλοι αναγνωρίζουν ότι ναι, ναι, μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα Ίσως δεν έχουν καταλάβει όλες τις δυνατότητες που το κείμενο προσφέρει. Ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η υλοποίηση γίνεται με ανοιχτό ευρύ πνεύμα, σε άλλες όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ για την ώρα δεν έχω διαπιστώσει κάποιο συγκεκριμένο σημαντικό μεγάλο πρακτικό πρόβλημα. Ζητούμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ναι, ε, ζητούμε περισσότερες ώρες διαθέσιμες ε, για να μπορούν οι άνθρωποι να ε, κάνουν την δουλειά τους. Ωραία, ναι, αλλά πραγματικά, εάν εσείς έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, πραγματικά θα ήθελα να το συζητήσω μαζί σας χωρίς κανένα πρόβλημα. Και αν υπάρχει πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα, είμαι βεβαιωτάτη ότι θα βρούμε και λύση. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε με τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Καλβέ ε, Σαμπον. Ε, Καλημέρα σας, αγαπητή κυρία. Χαίρομαι που σας ε, ε, βλέπω ε, εδώ έτοιμοι να απαντήσετε απέναντι σε αυτούς τους μη ε, ευρωβουλευτές. Εγώ θα σας μιλήσω γαλλικά παρότι έρχομαι από την Ισπανία. Τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά και άλλωστε τα αγγλικά δεν θα είναι πλέον κοινωτική γλώσσα οπότε δεν μας νοιάζουν κιόλας. Θέλω να σας υποβάλω τρία ερωτήματα. Έχω ε, στην χώρα μου την ε, Banco Popular και γι' αυτό θα ήθελα να σας μιλήσω. Πριν από ένα χρόνο, πριν από ένα χρόνο, χρόνο έγινε η διάσωση του Banco Popular. Επομένως, σας υποβάλλω το εξής ερώτημα. Δεν πιστεύετε ότι ένα χρηματοπιστωτικό ε, σύστημα χωρίς έναν δανειστή τελευταίας ευκαιρίας ε, δεν είναι βιώσιμο. Επίσης, δεν πιστεύετε ότι για να μην χρειαστεί να πουλήσουμε ε, ε, νύχτα και ερήμην όλων μια τράπεζα, αλλά να γίνει σωστά, δεν θα έπρεπε ο οργανισμός του οποίου προείσταστε να έχει κάποιες επιπλέον δυνατότητες έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνει τέτοιες διαδικασίες. Επόμενη ερώτηση. Ωραία, είπαμε για την Λετωνία. Η οργάνωσή σας, η υπηρεσία σας μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ε, ωραία, αλλά παρόλα αυτά είναι δυσάρεστο. Είναι δυσάρεστο λέω να ξέρουμε ότι τελικά οι Αμερικάνοι είναι αυτοί που μας ε, άνοιξαν τα μάτια και μας έβαλαν ψήλους στα αυτιά. δεν πρόκειται να έχουμε αξιόπιστη, ε, αξιόπιστο κοινό νόμισμα ε, για ολόκληρο τον κόσμο εάν ε, δεν έχουμε συνεργασία. Εάν δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις σωστές, τότε πάμε προς την καταστροφή. Πρέπει να έχουμε ένα ευρώ το οποίο δεν θα χρειάζεται διαρκώς να το εξαγοράζουμε να, ε, ή να αποδεικνύουμε την εμπιστοσύνη που το έχουμε κάθε, χρόνο, κάθε μήνα. Συγγνώμη. Επιτέλους, επιτέλους λέω, ε, λάβατε υπόψη ε, και τα όσα συνέβησαν στην Deutsche Bank Paribas. Όλα καλά. Αλλά ότι τα στοιχεία του ενεργητικού, ιδιαίτερως ε, του τομέα 3, ε, ε, αντιμετωπίζονται ισοδίκια και με τον ίδιο τρόπο παντού. Θα ζητήσετε σε ορισμένους να μειώσουν την συνεισφορά όσον αφορά κάποιες κατηγορίες έτσι ώστε να, είναι πιο αξιόπιστα τα stress tests. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω στα γαλλικά γιατί χρησιμοποίησατε τη μητρική μου γλώσσα. Και λέτε ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου πλέον ε, λένε συνεχώ τα ίδια και τα ίδια, ενώ συνήθω οι εποπτικέ αρχέ σε εμάς κατηγορούν ότι λέμε συνεχώ τα ίδια και τα ίδια. Τώρα, ο δανειστής ε, ε, τελευταία ευκαιρία Πρέπει να παρέμβει να σώσει την τράπεζα με πιο νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν και αποφασίστηκε και από αυτό το κοινοβούλιο για να δοθεί ένα τέλος στο bailout, να σώνονται οι τράπεζες με τα χρήματα των φορολογουμένων και να έχουμε κανονισμό bail-in, να μοιράζονται τις απώλειες οι επενδυτές επίσης, οι οποίοι έχουν ε, ε, κέρδη είχαν στο παρελθόν από τα μερίσματα και ούτω καθεξής. Άρα, η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί, εκτός και να αλλάξει ο νόμος. Και μάλιστα πιστεύω ότι λύθηκε το θέμα με το σωστό τρόπο νομοθετικά, γιατί είδαμε σε ορισμένες χώρες ότι στήχησε εξαιρετικά ακριβά στον εθνικό φορολογούμενο η διάσωση των τραπεζών και δεν είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να ε, το ξανακάνουμε. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι στη Μάλτα και στη Λετωνία οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, είναι παρόντες και ούτε τελικά ξεκίνησαν το πρόβλημα. Ναι, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση εμένα διότι είμαι Ευρωπαία και προτιμώ και το λέω δημοσίως ότι είμαι υπέρ μιας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής για να καταπολεμήσουμε το κίνδυνο νομοποίησης παράνομων εσόδων σε ό,τι αφορά τα στοιχεία ενεργητικού επίπεδου 3, που, των οποίων η αξία αποτιμάται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα και μοντέλα, όλα αυτά τα παρακολουθούμε εκ του τα εποπτεύουμε σε στενά, βλέπουμε τις διακοιμάνσεις αυτών των στοιχείων ενεργητικού και μετά από κάθε επιθεώρηση προκύπτουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε επαληθεύουμε την αξιοπιστία των μοντέλων που χρησιμοποιούμε για αυτές τις αξιολογήσεις και αποτιμήσεις. Αυτά έχουν να κάνουν με τον έλεγχο επιτόπου και αυτό αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του δεύτερου πυλώνα που έχουμε. Ότι ζητούμε δηλαδή αύξηση κεφαλαιακής επάρκειας, αύξηση της ρευστότητας, καλύτερη διοίκηση και διαχείριση από πλευράς ε, τραπεζών και ούτω καθεξής. Τώρα, είπατε για την Banco Popular, η οποία είναι G-SIB, δηλαδή Παγκοσμίω Συστημικό Σημαντική Τράπεζα. Global Systemically Important Bank. Πράγματι, αυτό περιπλέκει τα πράγματα, το ότι είναι συστημικό σημαντική και άρα είναι πολύ πιο δύσκολη η εξηγίαση και η διάσωση της τράπεζας αυτής και γι' αυτό έχουμε επιπρόσθετη προϋπόθεση για κεφαλαιακή επάρκεια για την εκάστοτε συστημικό σημαντική τράπεζα. Νομίζω ότι η απόφασή μας είναι αρκετά ολοκληρωμένη, ότι λύνουμε και ασχολούμαστε επαρκώς με όλες τις πτυχές αυτού του θέματος Σημειώνω ότι η Επιτροπή της Βασιλείας έχει υποβάλει συγκεκριμένε συστάσεις για την επανεξέταση των στοιχείων ενεργητικού του κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και δυστυχώς τα ευρωπαϊκά κείμενα θεωρούνται ως reporting, ως επιπρόσθετες πληροφορίες του επόπτη. Όμως όχι, πρέπει η Επιτροπή της Βασιλείας τη σύστασή της να την ενσωματώσουμε πλήρως και να την υιοθετήσουμε πλήρως και για την αποτίμηση του ενεργητικού και για την απέτηση ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων. Και το θέλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό και ελπίζω να υπάρξουν εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βεν Γκίκολντ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Καλώς ορίσατε κυρία Ντανιέλ Νουή. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας θέσω το θέμα του οικονομικού εγκλήματος, του χρηματοπιστωτικού εγκλήματος στο πλαίσιο της δικής μας Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Σας καλώ λοιπόν να αναπτύξετε αυτό το θέμα στο βαθμό που μπορείτε εδώ, να μας πείτε τι κάνατε από την τελευταία φορά που σας είδαμε. Τι έχετε κάνει έκτοτε. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Τι κάνατε και πέρα της γνωστής ε, υπόθεσης της τράπεζας ε, Πιλάτου στη Μάλτα. Καταλαβαίνω δεν μπορείτε να σχολιάσετε ε, κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει και άλλη τράπεζα, η Sata Bank, που αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένε κατηγορίες και έχει χρησιμοποιηθεί για να εξαπατήσει τους καταναλωτές. Η Μάλτα είναι μικρό μέρος και έχει 28 τράπεζες, ένα μικρό νησί. Είχαμε την τράπεζα Νεμέα, την τράπεζα Πιλάτους και μετά την Σάτα Μπάνκ. Δεν εξετάσατε ποτέ το ενδεχόμενο να ελέγξετε το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Μάλτας γιατί ελοχεύει κίνδυνος χρηματοπιστωτικού ή οικονομικού εγκλήματος. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν είναι μέρος της νομικής μου αρμοδιότητας η καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, το anti-money laundering. Συνεργάζομαι με τους συναδέλφους της Μάλτας και της Λετωνίας για να είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνουν πλήρως τις ευθύνες που φέρουν για αυτά τα ζητήματα, ότι ε, αυτό διακινδυνεύει τη φήμη του ESSM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ε, είναι μικρές χώρες, αν θέλουν ε, βοήθεια πρέπει να τη ζητήσουν και εμείς ευχαρίστως θα την προσφέρουμε. Τόσα μπορώ να κάνω. Γιατί δεν είναι βέβαια η περίπτωση του FBLV, αλλά οι, περισσότερε οι περισσότερες ε, τράπεζες από αυτές είναι μικρές τράπεζες, λιγότερο συστημικό σημαντικές τράπεζες που δεν εποπτεύουμε άμεσα εμείς οι ίδιοι και ακόμα και όταν τις εποπτεύουμε είναι αρκετά δύσκολο να ε, αναλάβουμε προληπτική δράση. Καταρχάς, Οποιαδήποτε πραγματική δράση με βάση την καταπολέμηση του ε, ξεπλήματος χρήματος πρέπει να βασίζεται σε εμπειρικά στοιχεία που έχει προσκομίσει η Εθνική Εποπτική Αρχή. Τώρα, οι περισσότερες από αυτές τις τράπεζες είναι αρκετά έξυπνες και δεν ε, τραβούν την προσοχή των εποπτικών αρχών. Μένουν εκτός ραντάρ, αν θέλετε, γιατί έχουν αρκετή κεφαλαϊκή επάρκεια, επαρκή ρευστότητα και στη βαθμολογία, αν έβαζε κανείς ένα μηχάνημα να δώσει βαθμολογίες, θα έδινε την υψηλότερη βαθμολογία σε αυτή τη τράπεζα. Έτσι δεν μας τραβούν την προσοχή. Άρα, τι πρέπει να γίνει. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πυλώνα 2 και μπορούμε να εξετάσουμε το επιχειρηματικό τους μοντέλο, ότι βασίζονται υπερβολικά πολύ σε εξωτερικούς πελάτες, σε ξένους πελάτες, έξωθεν προορμόμενους και προερχόμενους για παράδειγμα. Μπορούμε να ζητήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα στον πυλώνα 2, αλλά όχι και πάρα πολλά, γιατί ο δεύτερος πυλώνας αποτελεί μια απλή μικρή ε, προσθήκη από αυτά που προκύπτουν από την νομοθεσία του επίπεδου 1. Και έχουμε και την ίδια αξιολόγηση, δηλαδή το κατά πόσο η εθνική νομοθεσία μας επιτρέπει να δράσουμε. Υπάρχουν χώρες όπου άνθρωποι που δεν θεωρούνται σωστοί, να το πω έτσι, δεν μπορούν να εκδιωχθούν από τα διοικητικά συμβούλια μέχρι ότου τελεσίδικήσει η υπόθεσή τους σε τρίτο βαθμό, σε τελεσίδικο οριστικό βαθμό από τα εθνικά δικαστήρια. Τώρα, κατά τα λοιπά, μπορούμε να αποσύρουμε τις συμφωνίες που αποτελεί και την ύψιστη τιμωρία για μία τράπεζα, μόνο όμως επί τη βάση των στοιχείων που μας έχει παράσχει η Εθνική Εποπτική Αρχή. Άρα δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, δεν είμαστε καλά εξοπλισμένοι. Ορισμένες φορές η μέθοδος μας λειτουργεί, άλλες φορές όχι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Ματ Κάρτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίσατε κυρία Νουή. Θα ήθελα να στρέψω την προσοχή μου στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μας λέει ο κύριος Κάρθη. Παρακολούθησα τις ε, απαντήσεις που δώσατε στο γραπτό ερώτημα που σας είχα απευθύνει και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και θα ήθελα να σας καλέσω να επαναξετάσετε την πρόταση που σας έχει υποβάλει η Επιτροπή Οικονομικών του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου για να έρθετε στην Ιρλανδία και να συζητήσετε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την τραπεζική προστασία στην Ιρλανδία. Γιατί πιστεύω ότι ε, υποεκπροσωπούνται οι Ιρλανδοί ε, στο γραφείο σας και γενικά ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μιλούμε κυρίως για τα ενυπόθηκα δάνεια. Και οι απαντήσεις σας δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει εκφράσει καμία προτίμηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μειώσουν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων οι τράπεζες. Και τα προϊόντα split mortgage έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επαναταξινομηθεί μέρος του δανείου ως ε, ε, ε, εξυπηρετούμενο. Για το PTSB φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τα πρότυπα τα απαραίτητα. Και μιλούμε για bond sales ε, σε σχέση, ε, δηλαδή πωλήσει ομολόγων, ε, οι οποίες συνδέονται με την τιτλοποίηση ενυπόθηκων δανείων και κατοικιών και στεγαστικών δακείων. Υπάρχουν κίνδυνοι και για αυτούς που έχουν το δάνειο και το εξυπηρετούν, και για να υπάρξει, υπάρχει κίνδυνος να διαδοθεί κάθε απειλή και να μολύνει αν θέλετε και την υπόλοιπη οικονομία. Άρα πρέπει να προστατεύσετε τους καταναλωτές. Πρέπει να το λάβετε αυτό υπόψη σας και στην αναθεώρηση που θα προτείνετε για τις εποπτικές αρχές. Ευχαριστώ. Ναι, ξέρω ότι μου προσφέρθηκε δυνατότητα να επισκεφθώ την Ιρλανδία και να μιλήσω ενώπιον της Επιτροπής σας για το θέμα αυτό, όμως ε, η πρόσκληση ήρθε τελευταία στιγμή και οι μέρες που μου προτάθηκαν δεν μου επέτρεπαν αυτή την επίσκεψη. Τη μια μέρα ήμουν στην Ελλάδα, 15 Μαΐου, κάτι τέτοιο, έτσι τα λέω απ' έξω, αν τυχόν κάνω κάποιο λάθος ε, στις ε, ημερομηνίες, συγχωρήστε με. Πάντως είχα μια πρώτη πρόταση για την Ελλάδα, και μετά είχα και συμμετοχή σε επιτροπές προσλήψεων. Ήταν πολύ δύσκολο να το αλλάξω αυτό. Βέβαια, του τουλεχθέντος παρατήρησα και ότι ο Ιρλανδός που είναι μέλος στο Ποπτικό μας Συμβούλιο ήταν εκεί στην επιτροπή αυτή. Επομένως, υπήρχε η δυνατότητα να εξεταστεί να εξηγηθεί αυτή η κατάσταση και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εποπτεία. Αφού είμαστε σε απόλυτο συντονισμό για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η προληπτική αυτή παρακολούθηση με βάση και τις δικές μας συστάσεις. Επομένω, εγώ δεν θα είχα και πολλά να προσφέρω. Αυτό που θέλω όμως να υπενθυμίσω είναι αφενός μεν ότι δεν μπορώ να λάβω επιπλέον ρόλο για την προστασία των καταναλωτών διότι δεν έχω αρμοδιότητα νομικά Υπάρχει αρμόδια αρχή υπό την ε, Ιρλανδική Κεντρική Τράπεζα, αρμόδια για την προστασία των καταναλωτών. Το του λεχθέντος δεν ε, μιλούμε για εκποίηση των ε, μη εξυπηρετωμένων δανείων. Με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζονται αναλόγως του αν πρόκειται για μεγάλη εταιρεία, μικρομεσαία, ιδιώτη, ούτω καθεξής. Το θέμα αυτό όμως του διαχωρισμού των δανείων και η Άιλον το έχει εξετάσει και άλλες αρχές και νομίζω ότι μπορούν να δώσουν ικανοποιητικές λύσεις αναλόγως της κατάστασης. Νομίζω ότι μπορούμε έτσι να εξασφαλίσουμε ένα ποσοστό, μια διαφοροποίηση ανάλογα με το ποσοστό της ε, ε, κάλυψης του χρέους αυτού 50-60, πόσο μέρος εξυπηρετείται. Αλλά πάνω απ' όλα κοιτάμε πρώτα σε ποιο βαθμό είναι βιώσιμο για τον πελάτη. Και βέβαια αντίστοιχα το ε, επιτόκιο που καλύπτεται, ο βαθμός μαρών κάλυψης από τις εγγυήσεις και μετά υπάρχει και το άλλο κομμάτι εάν η τράπεζα διατηρεί το δάνειο αυτό μέχρι ότου αποπληρωθεί τελείως ή όχι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. και θεωρώ ότι προσφέρει μια αρκετά καλή και λογική λύση. Οι τράπεζες πρέπει να είναι πάντως προσεκτικές. ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται αυτά τα δάνεια για να μπορεί ο πελάτης να τα εξυπηρετήσει. Γιατί εάν δεν εξυπηρετούνται η τράπεζα θα φτωχύνει περισσότερο από ό,τι αν τα είχε κρατήσει. Αυτό μας το δίδαξε και η κρίση των subprimes της ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Μάρκο Βάλλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα δώσω στην ε, πρόεδρο το χρόνο να βάλει τα ακουστικά της. Λοιπόν, μετά όσα είδαμε πρόσφατα και τα στοιχεία που λάβαμε, οι δραστηριότητες δεύτερου και τρίτου επίπεδου των τραπεζών που είναι υπό ε, εποπτεία του SSM δείχνουν 3,43 και 189 δις ανάλογα στο τρίτο επίπεδο δραστηριοτήτων και 3,13 και 141 δις σε ποσά που έχουν συγκεντρωθεί σε γερμανικές και γαλλικές αντίστοιχα τράπεζες με τα τεστ αντοχής θα πρέπει να γίνει τώρα για πρώτη φορά ε, μια αξιολόγηση αυτού του ενεργητικού. Αν είναι ρευστοποιήσιμο, βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο να αξιολογηθεί αυτό και είναι πιο δύσκολο να εξεταστεί σε ποιο βαθμό μπορεί αυτό το, ενεργητικό, αυτό το παθητικό μάλλον να οδηγήσει σε συστημική κρίση. Μετά πρέπει να εξεταστούν τα εσωτερικά συστήματα που χρησιμοποιούν αυτές οι τράπεζες για να αξιολογήσουν την τιμή αυτών των ε, ενεργητικών. Επομένως είναι αρκετά πλήρη αυτά τα στοιχεία, αυτές οι μέθοδοι είναι πλήρης. Και θα ήθελα να μας ε, πείτε εσείς αλλά και το SSM πώς απαντάτε στους ε, αμφισβητείες, εκείνους που θα τον αναμφιβόλω την μεθοδολογία, την αξιοπιστία αυτών των μέσων αξιολόγησης της αξίας και πώς εκτιμάτε την, ε, τις κάποιες αδυναμίες ενδεχομένως των εσωτερικών συστημάτων. Έχετε κάποιο τρόπο δηλαδή να δοκιμάσετε τη στεναρότητα των εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης αξία του ενεργητικού. Απάντηση. Ναι, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς επιτρέψτε μου να απαντήσω ότι αυτό το ενεργητικό είτε επίπεδο 3 είτε επίπεδο 2 πρέπει να καλύπτεται και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης και κυρίως μετά την κρίση είναι σαφές πως οι μεγάλες εταιρείε χρειάζονται για τις εξαγωγές τους και για κάθε μορφή δραστηριότητα ανάπτυξής τους ενεργητικό που να μην είναι τοξικό, που να μην είναι μη εξυπηρετούμενο. Και άρα αυτό δεν πρέπει να το προσφέρουν οι τράπεζε. Αν θέλει ο νομοθέτη να σταματήσουν οι τράπεζε να διαθέτουν τοξικό ενεργητικό, θα πρέπει απλώ να νομοθετήσουν ότι απαγορεύεται. Αν και αυτό ήταν ε, λάθο κίνηση για μένα, γιατί και αυτά τα προϊόντα είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση της οικονομία. Η συγκέντρωσή τους βρίσκεται στις μεγάλες τράπεζες, ναι. Συμφωνώ με τα ποσά αλλά όντω μερικές φορές ξαφνιαζόμαστε όταν βλέπουμε και μεσαίου μεγέθου τράπεζε. Τι οποίε επίση παρακολουθούμε με την εποπτεία μας για τη δραστηριότητα που έχουν, ώστε ο έλεγχος του κινδύνου να είναι αντίστοιχος με το μέγεθος και την περιπλοκότητα των ε, συναλλαγών τους. Όλα αυτά εντάσσονται στα τεστ αντοχής Αλλά βεβαίως εμείς δεν καθορίζουμε τα σενάρια των τεστ αντοχής. Σε μεγάλο βαθμό αυτά τα ετοιμάζει το, συστημικό, ε, το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και τα ψηφίζει η ΕΜΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Εμείς δεν συμμετέχουμε εκεί. Άρα και αυτό είναι βέβαια καλό. Ακολουθούμε τα σενάρια όπως ο χρήστης ε, τα κρίνει σημαντικά ή σωστά και έτσι δεν έχουμε και ε, σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα ως προς την αξιολόγηση αυτού του ενεργητικού και την ικανότητα αξιολόγηση των μοντέλων. Σας βεβαιώ ότι έχουμε κατάλληλο προσωπικό, χωρίς να πω ότι είναι και πολυπληθές, πάντως έχουμε αρκετό κόσμο στις τάξεις μας με τις σχετικές γνώσεις σε συνεργασία με τον SSM επίσης μπορούμε να στενώσουμε τις δυνάμεις μας και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και διασυνοριακές ε, εποπτείες, αυτοψίες για την ακρίβεια. Ενεργητικό επίπεδο 2 και 3 δηλαδή των τραπεζών ε, ελέγχονται με αυτοψίες επιθεωρητών που έρχονται από άλλη χώρα και άρα δεν υπάρχει ζήτημα μεροληπτικής ε, αξιολόγησης και ταυτόχρονα μπορούμε να έχουμε και καλή κάλυψη γενικά του θέματος. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι εάν θέλετε να είμαστε ακόμη πιο ενεργοί ως προς την προαγωγή μιας καλύτερης νομοθεσίας ακόμη για τις συναλλαγές των τραπεζών, υπάρχει πρόταση από τη Βασιλεία προέρχεται, είναι επιτάπητος, δεν έχετε παρά να την εφαρμόσετε. Και πρέπει να εφαρμόσετε σωστά για την εποπτεία μας κύριος Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ, κύριε Κάπλ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Περιμένω για τα ακουστικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ που είσαστε εδώ, κύριε Νουή. Θα ήθελα να τοποθετηθώ σε ένα θέμα το οποίο και εσείς θίξατε στην αρχή της εισήγησής σας. Ο τεστ αντοχής του Μαΐου του 2018 και την κατάσταση των ε, πολλών συστημικών, ελληνικών συστημικών τραπεζών και τις ευκρινήσεις που δόθηκαν και τα αποτελέσματα τα οποία θα δημοσιευθούν σε ύστερο χρόνο. Δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητική ή ιδιαίτερα καλή η κατάσταση για τις συστημικές τράπεζες. Έχουμε δυσμενή οικονομικά σενάρια με απόλυση μέχρι 15,5 δισεκατομμυρίων με τη χειρότερη για την τράπεζα πυρός 14,8 και αντίστοιχα και άλλες τράπεζες αναμένεται να έχουν ένα ποσοστό μείωσης κεφαλαίου σε επίπεδο 3,5% κατά μέσο όρο. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αποδειχθεί ε, ανθεκτικό στην κρίση, χρειάζεται ανακεφαλαίωση, υπόθηκε και νωρίτερα αυτό. 23% των ε, δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα, είναι, είναι διπλάσιο το ποσοστό από ότι στις Ιταλικές τράπεζες, από αυτό που διακρατούν οι Ιταλικές τράπεζες που είναι στο 11%. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς κρίνεται την κατάσταση για τις ελληνικές τράπεζες μετά από τα, τα τέστα αντοχής και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με μια θηγατρική της Τράπεζας Πυραιός ε, και την ιδιωτικοποίηση σε σχέση με τη, με τη Βουλγαρική Τράπεζα. Και η Postbank, θηγατρική της ε, Deutsche Bank, ενδιαφέρονται για αυτή την ιδιωτικοποίηση. Επομένως, αυτή, αυτό το, το δίδυμο, η Deutsche Bank με την Postbank και η Πυραιός με την Βουλγαρική, ε, τι εικόνα δίνουν και πώς μπορεί να υπάρχει ζήτημα ή αν μπορεί να υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αν στενωθούν αυτά. Και βέβαια με την ανακεφαλίωση του 2015 μπορούμε να περιμένουμε ε, την ανάγκη για περιορισμό των δραστηριοτήτων των ελληνικών τραπεζών. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Κατανοώ ότι θεωρείτε ότι ε, μπορεί να υπάρχει μια μείωση 9% του CTN σε, μια, σε, μια, ε, σε ένα σενάριο αντίθετο ε, κακής κατάστασης για την Τράπεζα πηρεώσει για άλλες ελληνικές τράπεζες. Εγώ θα έλεγα ότι οι ελληνικές τράπεζες καλά τα κατάφεραν κατά τη διάρκεια των stress tests. Ε, έχουν βεβαίως ε, ζητήματα και προβλήματα, αλλά ακριβώς ε, επειδή έχουν μεγάλη έκθεση σε μια τέτοια άσκηση ε, όντως είχαν έλλειψη ε, ενεργητικού αλλά η ανακεφαλαίωση, η ανακεφαλαιοποίηση συγγνώμη, ε, ήταν ε, απαραίτητη αλλά για λόγους επιτυχούς προώθησης και όχι ως υποχρέωση και οπωσδήποτε υπάρχει ε, παρακολούθηση όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, ναι, είναι γεγονός ε, ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι τόσο υγιείς όσο θα θέλαμε να είναι ενδεχομένως, αλλά παρόλα αυτά καταβάλουν προσπάθειες, προοδεύουν προχωρούν ε, και η κυβέρνηση και οι ε, ρυθμιστικές αρχές ε, υποβοηθούν και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι τουλάχιστον ενθαρρυντικά, τα αποτελέσματα των stress tests των ελληνικών τραπεζών και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ε, ε, ε, πραγματικά αποτελεί ενθάρρυνση, ενθαρρυντικό στοιχείο έτσι ώστε να προχωρήσουμε, έτσι ώστε και το θέμα των μη εξυπηρετουμένων δανείων να αντιμετωπιστεί με ικανοποιητικό τρόπο, αυτά να μειωθούν κτλ. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δεν μπορώ να ε, σχολιάσω ε, για μεμονωμένες ε, τράπεζες. Εγώ ήθελα απλώς να πω ποια είναι η ευρύτερη εικόνα. του Ματουτσέλο. Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούνε οι πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις ε, χωρίς ε, να λάβουμε υπόψη μας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ποιοι άλλοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που βλέπετε εσείς στο τραπεζικό τομέα της Ευρώπης. Πιστεύετε ότι ε, για η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης με τον έντις είναι μια σωστή λύση. Δεύτερη ερώτηση. ορισμένος, όχι όλες οι τράπεζες στην Ιταλία, όμως όλες, ακόμα και οι πιο μικρές, χρησιμοποιούν το σύστημα IFRS. Επομένως η κατάσταση στην, Ευρώπη δεν είναι παρόμοια. Άλλες, ε, χρησιμοποιούν, άλλες όχι ε, τα συστήματα. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε μια ενοποιημένη βάση λογαριασμών. Τρίτον, η, σήμερα ε, το Οικονομικό Ινστιτούτο της Γερμανίας θεωρεί ότι από το 2,6 σε 2,8 θα είναι το ποσοστό αύξησης. Η οικονομία όμως ε, δεν ε, ε, έχει γενικά προχωρήσει θετικά και πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να χειροτερεύσει την κατάσταση των γερμανικών τραπεζών. Τελευταία ερώτηση. Μας διαβεβαιώνετε ότι στο τέλος της εντολής σας δεν θα εργαστείτε για, γαλλικές, για λογαριασμό γαλλικών τραπεζών. Θα αρχίσω από το τέλος. Δεν θα δουλέψω για γαλλικές τράπεζες. Έχω δεοντολογικούς κανόνες, ηθικούς κανόνες ε, ε, που με εμποδίζουν. Υπάρχουν άλλωστε οι κανόνε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και των Γαλλικών Τραπεζών. Ε, απ' την άλλη πλευρά δεν είμαι και νεαρή, ε, επομένω δεν νομίζω ότι έχω πολλά περιθώρια να ξεκινήσω μια δεύτερη καριέρα. Ε, ίσως ε, ε, θα πρέπει να αναλάβω πλέον τα καθήκοντα ως ε, γιαγιά. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω γιατί είμαι γεμάτη ενέργεια, είμαι δραστήριο άτομο και επομένως εκτός από το να ε, ασχοληθώ με τα εγγόνια μου, ε, προφανώς θα κάνω και κάτι άλλο, πάντως όχι δεν θα δουλέψω για γαλλικές τράπεζες. Ε, ποιες είναι οι άλλες ε, τράπεζες SSM, Τώρα, όσον αφορά τον κίνδυνο, νομίζω ότι ε, ο κίνδυνος για τις ευρωπαϊκές ε, τράπεζες ε, είναι το θέμα της αποδοτικότητας. Υπάρχουν τράπεζες οι οποίες δεν έχουν την απαραίτητη κερδοφορία και αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μια τράπεζα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κερδοφορία. Είμαστε 10 χρόνια μετά από την κρίση και επομένως πρέπει να καλύπτονται αυτές οι οικονομικές προϋποθέσεις. Ε, όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, ναι, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Ε, συχνά έχω παραθέσει την περίπτωση της Banco Popular που αν δεν είχε λυθεί με την βοήθεια της Banco Santander και αν δεν είχε βρεθεί οποιαδήποτε ε, λύση ε, τότε θα έπρεπε ε, να είχε βρεθεί κάποια θα έπρεπε να είχε διαλυθεί και αυτό θα είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στους Πορτογάλους λόγω του SSM τα πράγματα ε, μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρα και ούτως ή άλλως οπότε δεν ξεκινάμε ε, με μια λευκή ε, κόλλα και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, μηδενικός κίνδυνος σε όλες τις χώρες. Ναι, οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντική η μείωση του κινδύνου και είναι μια καλή συγκυρία για να ξεκινήσει η διαδικασία έντης και ασφάλισης και συνασφάλισης κλπ όντως, όντως Υπάρχουν κάποιες χώρες, υπάρχουν κάποιες τράπεζες μάλλον σε ορισμένες ε, χώρες οι οποίες ε, ε, δεν χρησιμοποιούν τις ενοποιημένες διαδικασίες. Τώρα εάν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς αυτή την κατάσταση, όχι. Γιατί οι νομοθέτες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχουν κάποια, κάποια γενικά λογιστικά πρότυπα, υπάρχει το IFRS και εμείς λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε Οπότε ε, υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Ελπίζω να σας στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Νόη. Νουή, λέει ο κύριος Φερνάντεθ. Θα σας κάνω τρεις ερωτήσεις για το κοινό σύστημα εγγύησης αποταμιεύσεων και καταθέσεων. Στην πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, περιλαμβάνει μια σειρά από αιρεσιμότητες για να υπαχθεί κανείς σε αυτό το καθεστώς και μάλιστα στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο τους τελευταίους μήνες έχει συζητηθεί το Banking Package ε, που θα ψηφίσουμε στη συνέχεια και την πρόταση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θεωρείται απαραίτητη την επιβολή επιπρόσθετων όρων και προϋποθέσεων για το κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Εάν τελικά καταλήξουμε να έχουμε κοινή εγγύηση καταθέσεων ή αποταμιεύσεων, το δικό σας θεσμικό όργανο από τη στιγμή που είναι εποπτικό συμβούλιο και εποπτεύει και ελέγχει την κατάσταση των τραπεζών, δεν θα αλλοιωθεί η δουλειά σας δεν θα είναι διευρυμένη εποπτεία από τη στιγμή που πρέπει να καλύψετε και τις ε, καταθέσεις. Σε ποιο βαθμό αυτό θα αλλοιώσει τη δουλειά σας και θα την αλλάξει. Έχετε τα μέσα για να φέρετε σε πέρα σε αυτό το καθήκον ε, εποπτείας και ελέγχου όταν ε, θα υπάρχει κοινό σύστημα εγγύησης από Και τρίτη ερώτηση, στο ίδιο πλαίσιο εποπτείας. Εάν μια τράπεζα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, εσείς μπορείτε να την αποκλείσετε από το Ταμείο για τη Διάσωση και Εξυγίαση των Τραπεζών, έτσι δεν είναι. Μπορείτε να πείτε ότι μια τράπεζα δεν μπορεί να χαίρει αυτού του καθεστώτος γιατί δεν συμμορφούνται με τις ε, προϋποθέσεις. Ή μπορείτε να υποχρεώσετε την τράπεζα να ε, συμμορφωθεί για να μπορεί να ε, συνεχίσει να εποφελείται από αυτό το Ταμείο για την Εξυγίαση και Διάσωση των Τραπεζών. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αιρεσιμότητα και τις επιπρόσθετες προϋποθέσεις για το κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, πιστεύουμε ότι πρέπει να οριστούν οι προϋποθέσεις οι επιπρόσθετες εκ των προτέρων, να είναι επαληθεύσιμες, να είναι ελέγξιμες, να είναι εφικτές και να συνδέονται νομικά με τις διάφορες φάσεις ε, της διαδικασίας, γιατί δεν είναι το ίδιο αν έχουμε αντασφάλιση και δεν είναι το ίδιο αν έχουμε άλλη ασφάλιση και το καθεξής. Και άρα δεν πρέπει να μεταφερθεί στο απότερο μέλλον το σύστημα αυτό. Τώρα, για τις ποιοτικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί επιτάπητος και ως προς την πρόοδο που θεωρούμε εμείς ότι χρειάζεται να σημειωθεί. Να αντιμετωπίσουμε τα ONDs που δεν συνοδεύονται από εγγύησει. Δεύτερον, να έχουμε εποπτεία των μεγαλύτερων τραπεζών και επενδυτικών επιχειρήσεων. Μιλούμε για τις τράπεζες που μετεγκαθίστανται από το Λονδίνο, οι επενδυτικές επιχειρήσεις. Να εναρμονίσουμε και να βελτιώσουμε τα εθνικά νομοθετικά συστήματα, να εναρμονίσουμε τις εποπτικές αρμοδιότητες για το fit and proper. Να διασφαλίσουμε ότι το καθεστώς παρεκκλήσεων, waiver, λειτουργεί σωστά. Το διασυναριακό waiver δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν υποβάλλουν αιτήσει να αποκτήσουν αυτό το waiver. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με την εθνική νομοθεσία. Στην αρχή της συζήτησης για το CRD5 και το CRR2 ε, υπήρχαν αυτά τα waiver τα διασυνοριακά, αλλά έχουν, έχουν αποσυρθεί η πρόοδος αυτούς τους πέντε τομείς θα είναι σημαντική και θα εξαρτήσουμε τη θέση μας από το πόσο ε, σημειώνεται πρόοδος για αυτά τα θέματα. Έτσι θα έχουμε μείωση κινδύνου και έτσι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο για την ε, ατζέντα την πολιτική του διαμοιρασμού του κινδύνου. Τώρα, αν ε, θα έχουμε εποπτικό ρόλο. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς, πολλές και διαφορετικές εποπτικές αρχές που να εποπτεύουν την κατάσταση με το κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Και οι εξουσίες και αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα. Έχει γίνει συζήτηση και γι' αυτό. Είναι σημαντική η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για το επίπεδο 3, για το Level 3 Regulation, Εμείς ε, είμαστε παρόντες και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε για το επίπεδο 1 και το επίπεδο 2. Μιλούμε για στενή συνεργασία. Αυτό είναι το διαδεδομένο ευρωπαϊκό μοντέλο μεταξύ των εποπτικών αρχών και του κοινού συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη εγγύηση για το ότι θα εκπληρώσουμε ε, τις υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις μας χωρίς να έχουμε επικαλύψεις. Τώρα, αν θα μπορέσουμε να αποκλείσουμε τράπεζες, δεν, το νομίζω. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουν και να το συζητήσουν αυτό οι νομοθέτες. Νομίζω ότι τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων πρέπει να συνενωθούν και τα σημαντικά τραπεζικά ιδρύματα που εποπτεύουμε και τα λιγότερο σημαντικά. τα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν υποβληθεί σε πλήρη αξιολόγηση. Ξέρουμε πολύ καλά τα δυνατά και τα αδύναμά του σημεία, αλλά αυτά θα αποφασιστούν με το Κοινοβούλιο. Από το Κοινοβούλιο, κατά πόσο χρειάζεται ε, πλήρης αξιολόγηση των λιγότερο σημαντικών συστημικών τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε εμείς την αρμοδιότητα να το κάνουμε αυτό και δεν θα το κάνουμε για να αποκλείσουμε τις τράπεζες. Καμία τράπεζα δεν αποκλείστηκε από το ε, εποπτεία του ESSM. Εκεί όπου χρειάζεται ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να λάβει χώρα. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Μετά είναι ένα καινούργιο σύστημα και πρέπει οι τραπεζικοί φορείς να είναι έτοιμοι για να μπορεί να υπάρξει κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Ευχαριστώ. Έχουμε καθυστερήσει. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους, ε, λέει ο πρόεδρος, οι συνάδελφοι να ε, κάνουν ερωτήσεις όχι παραπάνω από δύο λεπτά ο καθένας και η κυρία Νουή να απαντάει σε τρία λεπτά το περισσότερο. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ανταλλαγή αυτή απόψεων σήμερα. Δύο σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ στη συζήτηση μαζί σας. Το πρώτο έχει να κάνει με τις κυβερνοαπειλές, καθώς όλο και περισσότερο τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εν γέννη γίνονται στόχοι πολυαριθμών κυβερνοεπιθέσεων. Οι τράπεζε και τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ω εκ τούτου έχουν εγκαθιδρύσει μια σειρά από συστήματα προστασία. Θα ήθελα λοιπόν να ενημερωθώ για το πώς το SSM ε, συνεργάζεται με τις τράπεζες στην καθημερινή δουλειά της εποπτείας που έχει για τον περιορισμό αυτού του κινδύνου και εάν έχετε αναπτύξει συγκεκριμένε συστάσεις προς τις τράπεζες για το θέμα αυτό. Και επίσης, εάν θεωρείτε ότι οι τράπεζες της FinTech είναι πιο ευάλωτες στο κίνδυνο. Δεύτερον, κρατικό χρέος. Η κρίση κρατικού χρέους στην Ευρώπη έδειξε ότι ενεργητικό δεν μπορεί να θεωρηθεί επουδενή και ποτέ ε, άμυρο κινδύνου. Αυτή τη στιγμή έχουν ε, οι τράπεζες σημαντικό, διακρατούν σημαντικό ποσοστό και όγκο εθνικών χρεών που άρα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητά τους. Καταθέτει λοιπόν μια νομοθετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ε, τίτλους, κρατικά ομόλογα, αν και κάποια κράτη-μέλη φαίνεται πως έχουν κάποιους δισταγμούς για τις προτάσεις αυτές, θα ήθελα τη δική σας γνώμη. Ευχαριστώ. Απάντηση στα γαλλικά. Ε, αν μου επιτρέπετε, θα μιλήσω αγγλικά για να... Εκτός και να μου ζητήσετε να τα πω στα γαλλικά για να με καταλάβετε καλύτερα. Και στα αγγλικά κίνδυνος είναι όντως ε, κάτι πολύ δύσκολο για όλους τους οικονομικούς ε, παράγοντες, περισσότερο βέβαια για τις τράπεζες, όσο περισσότερη τεχνολογία πληροφορίας χρησιμοποιούν και μάλιστα απόρριτη ε, ενοποιημένη, κατανεμημένη καλύτερα, ε, τόσο πιο πολύ εκτίθενται στις κυβερνοεπιθέσεις. είναι κομμάτι της εποπτείας μας σε σχέση με τους λειτουργικούς κινδύνους ή εξετάση του κυβερνού κινδύνου. Σε σχέση με αντίστοιχους κινδύνους ε, έχουμε και εδώ ε, συγκεκριμένα εργαλεία. Στηριζόμαστε στην καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ακτιωτικής του 2017 για την εποπτεία της ε, πληροφορικής. Πολύ καλές κατευθυντήριες γραμμές και χρήσιμες που κυρίως τώρα αξιοποιούμε για την, ε, για την ε, αναγωγή στο cloud και περιμένουμε βέβαια και διευκρινήσεις από την έμπαση ως σημεία. Έχουμε αυτοψίες. Από την κοινή υποπτική ομάδα στα γραφεία. Αφενός, αφετέρου όμως έχουμε και τις αυτοψίες με αποστολές που έχουν στόχο να εξετάσουν τη διακυβέρνηση, την εξωτερική ανάθεση, την ασφάλεια, την συνέχιση, τη διαχείριση, την κυβερνοασφάλεια στην ηλεκτρονική, στις ηλεκτρονικές λειτουργίες. Και έχουμε ταυτόχρονα και ε, εγκάρσια θεματικές ε, μελέτες που αφορούν την κυβερνοασφάλεια το 2015 συγκεκριμένα, το 2016 εξωτερική ανάθεση στο cloud computing, στο νέφος δηλαδή. Τώρα η τελευταία έκθεση αφορά το, πιο γενικά τον, κίνδυνο, τον κυβερνό κίνδυνο για την πληροφορική. Χρησιμοποιούμε διάφορες πηγές ε, ενημέρωσης. Είχαμε παραδείγματι πέρσι υποχρεωτική καταγραφή επεισοδίων επιθέσεων ενώ τώρα ακολουθούμε τις, ε, τα δεδομένα τα, της αγοράς για την ε, έκθεση των τραπεζών στον κυβερνοκίνδυνο. Αλλά βέβαια δεν σταματάνε εδώ οι δράσεις μας. Όπως είπα και πριν, Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει ό,τι χρειάζεται. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Για τα ευρωπαϊκά ασφαλή ομόλογα. Safe points. Και γενικά ασφαλή, ασφαλείς τίτλους. Εξετάζουμε τις που τους καλύπτουν τους τίτλους αυτούς. Υπάρχει πρόταση της Επιτροπής ε, για την ρύθμισή τους, που είναι μια καλή κίνηση και οπωσδήποτε την υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Φροντζουλίτσα. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Ε, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή προσέγγιση η αναθεώρηση ε, της ε, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων ίσως να μην είναι αρκετή έτσι ώστε να επιτευχθεί η αρμονική συνεργασία γιατί δεν αφορά μονάχα τον εποπτικό προληπτικό έλεγχο το θέμα αυτό αλλά και την ποινική συνεργασία, συνεργασία για ποινικά θέματα. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες να συνεργαστούν. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι η πέπτη οδηγία ε, που εγκρίθηκε ε, από το Κοινοβούλιο πριν από λίγο καιρό ε, έχει, περιέχει κάποιους περιορισμούς όσον αφορά το απόρριτο που δυσκολεύει τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των προοπτικών αρχών και των αρχών. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι όσον αφορά το θέμα του ξεπλήματος χρήματος θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη συνεργασία. Δεύτερη ερώτηση. Λαμβάνοντα υπόψη ότι η ανταλλαγή απορρίτων πληροφοριών έτσι όπω ε, ε, προβλέπεται από την πέμπτη οδηγία δεν σημαίνει ότι οι αντίστοιχε αρχέ ε, θα συμμερίζονται εν ευθέτω χρόνο και σε δόκιμο μάλλον χρόνο όλε τι πληροφορίε. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιε σημαντικέ βελτιώσει που μπορούν να υπάρξουν έτσι ώστε να βελτιωθεί το ε, πρόγραμμα συνεργασία και το πλαίσιο ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Ευχαριστώ. Ε, θα απαντήσω στα αγγλικά εάν μου επιτρέπετε ή μήπω προτιμάτε στα γαλλικά. Ε, προτιμώ στα γαλλικά και να σας, απαντήσω γαλλικά. Εγώ προσπαθώ να βρω τον καλύτερο τρόπο έτσι ώστε να με καταλάβουν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι, λέει ο Μιλήτρια. Ε, με ρωτάτε αν πιστεύω ότι η πέμπτη οδηγία η οποία αναφέρει κάποια ενδεχόμενα μη δυνατότητα ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών, ε, ναι, ε, έτσι είναι, όμως είναι οδηγία, δεν είναι κανονισμός θα μεταφερθεί στην ε, νομική, ε, στο, στο νομοθετικό πλωστάσιο των 19 ε, χωρών, αλλά καταλαβαίνετε ότι η ενσωμάτωση παίρνει χρόνο. Δεν ξέρω για την προκειμένη περίπτωση, αλλά συνήθως είναι 18 μήνες, 20 μήνες, κάτι τέτοιο ε, για την ενσωμάτωση. Επομένως, για αρκετούς μήνες ακόμα, για αρκετό καιρό, θα ζούμε, αν θέλετε, με τις παλαιές διατάξεις, ε, όπου κάποιες χώρες, βάσει της εθνικής νομοθεσίας τους, μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μαζί μας, άλλες όμως δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Επομένως, η βελτίωση, κατά την άποψή μου, πρώτα θα προέλθει από, ευρωπαϊκή, ε, από ευρωπαϊκό κανονισμό και όχι ε, ε, ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκή οδηγία. Το άλλο ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία, η οποία ελέγχει την ορθότητα της εφαρμογή στι διάφορες χώρες και τη ενσωμάτωση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική έτσι ώστε να ε, είναι βέβαιο ότι η ενσωμάτωση γίνεται με τον σωστό τρόπο. Είναι γεγονός ότι και η εμπειρία και η τεχνογνωσία των διαφόρων χωρών δεν είναι παρόμοια. Ανέφερα προηγουμένως ότι η περίπτωση της Λετωνία είναι μια μικρή χώρα με μια ε, εποπτική αρχή που έχει περιορισμένο αριθμό προσωπικό, κάνουν ό,τι μπορούν φυσικά αλλά, αλλά, αλλά δεν έχουν απαραίτητα όλο τον εξοπλισμό, δεν έχουν απαραίτητα όλες τις δυνατότητες έτσι ώστε ε, να αντιμετωπίσουν μέτρα νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων τα οποία είναι πολύ προχωρημένα και τα οποία ε, ε, εφαρμόζονται από ανθρώπους που έχουν μεγάλη εμπειρία γι' αυτά. Επομένως, ο SSM ε, ή μια τέτοια αντίστοιχη μορφή για τις συνεργατικές τράπεζες οπωσδήποτε θα πρέπει να προβλεφθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κύρτσος. Ε, thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα υποβάλω ερωτήσεις ε, στα ελληνικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Με τα στοιχεία, οι ελληνικές τράπεζες πηγαίνουν καλύτερα, συμφωνώ και με την εκτίμηση της κυρίας Νουή, και πέρασαν και τα λεγόμενα stress tests Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο προβληματίζει πολλούς αναλυτές, δηλαδή μεγάλος, μεγάλο μέρος των ιδίων κεφαλαίων τους είναι ο λεγόμενος αναβαλόμενος φόρος, δηλαδή το δικαίωμά τους να μην πληρώνουν φόρους τα επόμενα χρόνια και φυσικά ε, με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται τα ίδια κεφάλαια. Ε, ανησυχεί την κυρία Νουή αυτό το θέμα και δεν κάνω κριτική γιατί και η κυβέρνηση το ψήφισε και το κόμμα μου που είμαστε στην αντιπολίτευση το ψήφισε αλλά αναρωτιέμαι σε οικονομικό επίπεδο ε, είναι καλό για τη σταθερότητα των τραπεζών. Κερδίζουμε χρόνο, θα πάμε σε κάποιες επόμενες δυσκολίες. Τι ακριβώς γίνεται. Και η δεύτερη ερώτηση έχει σχέση με, τις, ε, με τους πληστηριασμούς ακινήτων, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει σε αρκετά μεγάλη κλίμακα. Αυτό είναι δύσκολο αλλά αναγκαίο, όλοι το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει όμως το εξή Από τα ακίνητα που πολλούνται, που πουλάνε οι τράπεζες, τελικά ένα 80 με 90% καταλήγει στις ίδιες τράπεζες. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλοι αγοραστές να ενδιαφερθούν. Ε, σας προβληματίζει αυτό. Δύο τεχνικές θα έλεγα ερωτήσεις που μπορεί να έχουν σημασία. Ευχαριστώ. Thank you very much uh, for your question. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας. Δεν είναι και πολυτεχνικά. Το πρώτο για τον αναβαλλόμενο φόρο έχει να κάνει με την ποιότητα της κεφαλαιακής επάρκειας και τη δυνατότητα του κεφαλαίου να απορροφήσει τις απώλειας. Τις απώλειες. Μου αρέσει ο αναβαλλόμενος φόρος? Όχι, δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει αυτό. Είμαστε στη φάση του phasing out, της σταδιακής εξάλληψης αυτής της δυνατότητας. Και τελικά θα ολοκληρωθεί η φάση του phasing in της σταδιακής εισαγωγής και θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα στοιχεία ενεργητικού με διαφορετικό τρόπο. Δεν το κάνουν όμως μόνο οι ελληνικές τράπεζες. Δεν είναι η κατάσταση πολύ διαφορετική στις ελληνικές τράπεζες από ό,τι σε άλλες μη ελληνικές. Τώρα για το δεύτερο σας ερώτημα, για τους πληστηριασμούς, είναι σημαντική για τα μεγάλα κίνητα υψηλή αξίας, γιατί υπάρχουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, ζώμενοι που θα μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνειά τους, αλλά δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν κι άλλοι. Άρα δεν βλέπουν κανένα λόγο να ξεπληρώσουν το χρέος τους. και βλέπουν τα κίνητά τους να είναι στον κατάλογο με τους μελλοντικού πληστηριασμούς. Και όταν τα δουν αυτό να συμβαίνει, ε, τότε συνομιλούν με τις τράπεζες και βλέπουν τι μπορούν να κάνουν με αυτό το δάνειο, το να ρυθμιστεί για να γίνει εξυπηρετούμενο. Τώρα, είναι πρόβλημα το ότι οι τράπεζες ε, αποκτούν τα ακίνητα οι ίδιες και τα αγοράζουν οι ίδιες. Ναι, είναι πρόβλημα. Δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά Έχουμε τα foreclosed assets. Εάν η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ε, επιτυγχάνεται με ε, foreclosed assets, με ακίνητα που έχουν κατασχεθεί, τότε δεν μειώνεται η έκθεσή τους, δηλαδή δεν μπαίνει στο πυλώνα 2. Εξαρτάται βέβαια και ποια έχει κατάσχει. Κάποια στοιχεία ενεργητικού που έχουν κατασχεθεί από την τράπεζα έχουν αξία στην αγορά και το και δεν θέλουμε τελικά να τα θέσουν στην αγορά όλα μαζικά και να πέσει η τιμή τους και γι' αυτό θέλουμε να τα διακρατήσουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τώρα θα χρειαστεί χρόνος να αριθμιστούν όλα αυτά, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη η αξία αυτών των ακινήτων τελικά που διακατέχουν οι τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πολύ επικοδομητική αυτή ακρόαση. Η επόμενη θα λάβει χώρα στις 20 Νοεμβρίου. Πέντε λεπτά διάλειμμα πριν την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Να ξαναρχίσουμε λοιπόν. Ε, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια όσον αφορά την συνεδρία των συντονιστών. Ε, έχουμε EMF και σοσιαλιστές ε, την, την απονομή των, των πόντων. Επίσης ε, έχουμε για την ALDE ε, cover bonds, επίσης ε, έκθεση σε cover bonds, επίσης διασυνοριακή κλπ. Ελάχιστη κάλυψη για, το, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Εταιρική φορολόγηση για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ε, ε, οι χρεώσεις στις διασυνοριακές ε, διαδικασίες ΕΛΚ, τροποποίηση οδηγίας για το Λουγκάνο, ε, ΕΛΚ, ε, τίτλοι ε, και S&D, βιώσιμη ανάπτυξη πράσινη, τροποποίηση για τον κανονισμό για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος η ίδια ομάδα. E ECR για εγκληματικές ε, πράξεις, προστασία ε, των καταγγελόντων για ε, απάτες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΓΚΟΕ, ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η ΑΛΤΕ, ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του έτους η ΕΝΕΦ, η ΓΚΟΕ για την φορολόγηση των εταιριών, κατάσταση ε, του, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το ΕΛΚ. Το Προεδρείο θα κάνει ορισμένα ε, πράγματα επίσης. Για τον Ιούλιο θα έχουμε τον διοδομημένο διάλογο με τον Επίτροπο Κατάινεν διευκρίνηση ότι χρειάζεται ε, μία νέα ε, διοίκηση για την ΕΜΣΑ. Επίσης, ε, τον Ιούλιο θα έχουμε τα benchmarks. Δεν υπάρχει αντίρρηση όσον αφορά την μελέτη για, τις, για τους λογιστικούς ελέγχους. Επίσης για το SRSP Όλα αυτά λοιπόν τα είπαμε και μπορώ να σας ε, ζητήσω να κάνετε έναν έλεγχο. Ε, εν τω μεταξύ οι διερμηνείς ε, σας ενημερώνουν ότι βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω της εργασιακής διάνεξης με τη διοίκηση για τις συνθήκες εργασίας μας. Σε ορισμένες καμπίνες έχουν επιστατρευτεί όλοι οι διερμηνείς και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Αυτό ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμά του στην απεργία και συνιστά διάκριση προς τις υπόλοιπες γλώσσες. Ως εκ τούτου και σε ένδειξη αλληλεγγύης η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει στη στάση εργασίας που προβλεπόταν για τη σημερινή συνεδρίαση. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο έλεγχος και θα ξεκινήσουμε τώρα με την πρώτη ε, έκθεση Γκούναρ Χόκμαρ, SRMR.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 κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εναλλακτική συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική στην επόμενη σελίδα, η συμβαστική γ, σι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και είναι ισοπαλία 28 υπέρ 28 κατά επομένως απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 και 173 από ό,τι καταλαβαίνω από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Όχι. Πάρα πολύ ωραία. 177 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επομένως, ε, τροπολογία 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές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 αποχές απορρίπτεται. Ψηφοφορία επί της τροποποιημένης προτάσεως της Κομισιόν Διονομαστικής Κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 38 ψήφοι υπέρ, 8 κατά, 11 ε, αποχές, συγχαρητήρια στον εισηγητή και ε, ψηφίζουμε ε, τώρα για την πάλι με ονομαστική ψηφοφορία ε, την έναρξη πραγματεύσεων, άρχεται η ψηφοφορία. Ακόμα ένας άνθρωπος που πρέπει να ψηφίσουν. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. 39 ψήφοι υπέρ, 8 ψήφοι κατά, 10 αποχές. Επομένως θα ε, ε, ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις μετά από τις ε, σχετικές ανακοινώσεις στην Ολομέλεια. Δεύτερη έκθεση του εισηγητού Γκούναρ Χόκμαρ. Τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 71 όχι. Γιατί 70 έχει καταπέσει. Στην 71 υπέρ κατά αποχές Απερίφθη. Συμβαστική α υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρκατα κατά αποχές απερίφθη. 72 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 82 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 83 υπέρκατα... κατά Επαληθεύουμε τον 83 παρακαλώ. Αρχίζει. πέρας και απερίφθη. 94 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 84 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 84 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 86 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 88 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 89 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 90 υπέρ κατά α, περίφθη, 91 υπέρ κατά αποχές απερίφθη υπέρ αποχές απερίφθη, 93 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, υπέρ αποχές απερίφθη, 96 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, απερίφθη 97 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 98 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 99 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 100 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 101 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 102 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 103 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 104 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 105 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 106 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 107 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 108 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 110 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 109 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 111 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 112 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 113 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 114 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη 115 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε. 115. Πέρας. Και απερίφθη. 116 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 117 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 118 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 119 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 120 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 121 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη ε, 22, 23, 24 και 25 διαγραφές ταυτόσημα υπέρ κατά αποχές και εγκρίνονται. Καταπίπτουν οι λοιπές έως την 129 και πάμε στην 130. Όλες οι άλλες θα ήταν ταυτόσημες. 130 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 131 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 165 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 166 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 167 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 168 υπέρ κατά, υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 169 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 170 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 171 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 172 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 173 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 174 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική σύ με προφορική τροπολογία είναι προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Υπέρ. 176. Κατά. Αποχές απερίφθη, 177 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 178. Συμφωνούμε. 181 πήγαμε, 182 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε την 182. Ωραία, πέρας λοιπόν. 183 υπέρ εγκρίθηκε αυτό. 183 υπέρ. Επαληθεύουμε την 183. Πέρας. Πέρας και απερίφθη. 184. 184. Ψηφίζουμε 185 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά και επαληθεύουμε την 187. Πέρας. Εγκρίνεται 188 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη. 188. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ και ας συγκεντρωθούμε λίγο σε επαληθεύσεις έτσι να γίνονται επαληθεύσεις μόνο όταν είναι ανάγκη. 189 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη, 190 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. συμβαστική D δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εναλλακτική ε συμβαστική υπέρ κατά αποχές απερίφθη, συμβαστική ε να επαληθεύσουμε την εναλλακτική ε πρώτα πέρας 38 κατά 18 υπέρ απερίφθη. Συμβαστική ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Την ε θέλετε τη συμβαστική ε, μένει σε σαφές το αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, επαληθεύουμε. Έκλειση σας απευθύνω. Πέρασε και εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G, Z, πολλές σελίδες θα γυρίσετε για να φτάσετε εκεί. Κάπου στην 31 πέφτει, ανάλογα σε ποια γλώσσα το έχετε ίσως. Στην 31 στο δικό μου κείμενο, συμβαστική G. Υπέρ, είστε έτοιμοι για την G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται H ήτα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 413 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική ΑΙ δηλαδή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 485 Στη σελίδα 44 θα τη βρείτε, τουλάχιστον αυτό λέει ο δικός μου κατάλογος. 485 υπέρ κατά αποχές και απερίφθη. Ή 20 τώρα υπέρ κατά απερίφθη. Νομίζω ότι είναι σε σαφές, αλλά σε απολυθεύσουμε αν το θέλετε. Α, ναι, απολυθεύουμε. 20, τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Και απερίφθη. J υπέρ κατά από αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική K κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 505 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 508 υπέρ κατά επαληθεύουμε 508 παρακαλώ Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. Συμβαστική L λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 547. 547 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 548 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 549 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 550 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 551 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 564 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 565 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 566 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 567 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, Μετά, μετά. 568 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 569 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 570 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 571 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 572 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 573 υπέρ κατά απερίφθη νομίζω, αλλά δεν σηκώνεται και τα χέρια. Επαληθεύουμε. 573. Πέρας. Και απερίφθη. Αν block. Από την 574 ομού έως και την 577. Υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 578 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 30 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 32 υπέρ κατά υπέρ αποχές εγκρίνεται, 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 35 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, υπαριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 36, 36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 38 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 39 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 40 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 42 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 41 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 44 και 5. 44 και 5 προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 60 και 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία έτσι όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θέλετε να ελέγξουμε την 68? Ναι. Α, γιατί το ΕΛΚ ήταν υπέρ. Συγγνώμη. Σωστά. Άρα ψηφίζουμε την 68 α, ε, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 68. Ποιος είναι υπέρ. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι το ΕΛΚ ήταν κατά. Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 38 υπέρ, 14 κατά, 5 αποχές. Ψηφίζουμε την απόφαση να μπούμε σε τριμερή διάλογο. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 37 υπέρ. 14 κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια. Αξίζει το χειροκρότημα. Ο εισηγητής, η σκιώδης, η σύμβουλη, η γραμματεία. Εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ όλους. Προχωρούμε στην έκθεση Ζήμεν. Και ξεκινούμε με το CRD το 5. Μισό λεπτό. Συμβιβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική κάπα αλφα νέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συ, τροπολογία 103 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Για το φύλλο. Κάποιοι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμα ψηφίσει. Το κατόφλι είναι 13 μέλη για να ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 1.04 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμπιβαστική λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1.65 και 1,66 και 1,67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1,68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1,69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1,70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1,71 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. The vote is Πέρα εγκρίνεται με πλειοψηφία μίας ψήφου, 29 υπέρ, 28 κατά, 1,72 υπέρ. Α, ονομαστική ψηφοφορία, την 172. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 172. Vote is closed. Is adopted εγκρίνεται. 30 υπέρ, 28 κατά, 0 αποχές. 173 υπέρ, κατά. Την παληθεύουμε ηλεκτρονικά την 173. Πέρασε. Απορρίπτεται. 1,74. Υπέρ. Κατά με ίδια πλειοψηφία, αλλά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 174. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε, R. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην 188. Υπέρ. 188, 189 και 190 τις ψηφίζουμε μαζί αυτές τις τρεις υπέρ, κατά να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτονται, αλλά να το δούμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 31 κατά, 27 υπέρ. Πάμε στην 190. Υπέρ, κατά, άποχες, το επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 190. Πέρασα. Απορρίπτεται. 31 ψήφοι κατά 27 υπέρ. Συμβιβαστική μη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική μη ε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 199 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική νη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 31 ψήφοι υπέρ, 27 κατά. Τροπολογία 18 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.11. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 211. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.10. Υπέρ. Κατά. Νομίζω με την ίδια πλειοψηφία θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Γιατί θα μου το ζητήσετε, το ξέρω. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 29 υπέρ, 27, 29 κατά, 27 υπέρ, μία αποχή. 2-12 υπέρ. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 212, παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 31 ψήφοι κατά, 27 υπέρ. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική αλφα ε υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F και FA. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H. Όμως υπάρχει έτοιμο ονομαστικής ψηφοφορίας. Όχι, όχι. Πάμε στη συμβιβαστική H, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τη Ι συμβιβαστική, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 327, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.28 και 3.29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται, συμβιβαστική P, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, J επίσης εγκρίνεται, Προφορική τροπολογία υπέρ, κατά. Το ΕΛΚ είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3.38 υπέρ, κατά, να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 338. Παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Συμβιβαστική ΒΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΒΒ υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τη συμβιβαστική ΒΒ. Παρακαλώ πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Επομένως, τροπολογία 34 υπέρ, κατά. Ε, παρακαλώ πολύ να ψηφίσετε κανονικά, αλλά για την 34 θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ακόμα ε, δεν έχουν ψηφίσει όλοι οι συνάδελφοι για την τροπολογία 34. Πέρασε της ψηφοφορίας και απερίφθη η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 δεν ψηφίζεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική ε, ζήτηση ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική σι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβιβαστική σι μπι υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για, για την συμβαστική CB άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία 29 ψήφοι υπέρ 29 κατά, άρα πρέπει να, να ψηφίσουμε την τροπολογία 37 υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 37, δεν σηκώνετε τα χέρια σας δεν ξέρω τι έχετε ψηφίσει λέει ο Πρόεδρος, τροπολογία 37. Πέρας της ψηφοφορίας και απεορίπτεται τροπολογία 41 υπέρ ή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική C α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 379 όχι όχι λέει ο πρόεδρος αυτή Α, πρέπει να την ψηφίσουμε. Ωραία. 3,79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά η ηλεκτρονική υπαλήθευση για την τροπολογία 45 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται όμως. 46 ε, υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 46 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 47 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 47 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται Τροπολογία 421 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική SR υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 424 25, 427 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 51 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 53 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ υπέρ για την τροπολογία 5 Ψηφίστε παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 55 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτει την τροπολογία αυτή. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 58 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται τροπολογία 59 υπέρ. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, ψηφίζουμε την ε, τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. πέρα της ψηφοφορίας, 44 ψήφοι υπέρ, 4, ε, συγγνώμη, 5 ε, ψήφοι κατά, 8 αποχές ε, ψηφοφορία της αποφάσεως ε, για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων. Πάλι με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Το ψήφισμα θα το ψηφίσουμε άλλη φορά. Πέρας της ψηφοφορίας, 47 ψήφοι υπέρ 9 αρνητικές δύο αποχές. Και επομένως εγκρίνεται η απόφαση. Συγχαρητήρια κύριε Ισηγητά, αλλά θα χειροκροτήσουμε όταν θα γίνει η τελική ψηφοφορία και για το CRR2, ε, συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 2.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.34 υπέρ κατά παρακαλώ να ψηφίζετε με πιο ε, ορατό τρόπο. Για την ώρα κάνουμε ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για αυτή την τροπολογία. Πέρας. 25 ε, ψήφοι υπέρ, 28 ψήφοι κατά, επομένως δεν γίνεται δεκτή. Συμβιβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία F έχει γίνει δεκτή και επομένως φτάνουμε κατευθείαν στην τροπολογία Z Υπερκατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική και υπέρκαταποχέ αποχές εγκρίνεται, G υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 303 υπερκατά αποχές απορρίπτεται, 304 υπερκατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική ME υπερκατά αποχές εγκρίνεται. και περνάμε επομένως στην προφορική τροπολογία ε, επί του άρθρου 14 του εισηγητού υπερκατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 311 υπερκατά αποχές απορρίπτεται 312 υπερκατά αποχές εγκρίνεται 41 ζητώ συγγνώμη 41 καταπίκτη 314 υπέρ κατά αποχές, 314 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ελέγχουμε το αποτέλεσμα για την 314. Πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη η τροπολογία αυτή. 316 υπέρ, 316 υπέρ κατά Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση 316 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απερίφθη η συμβιβαστική CG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 325 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, σε AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AK υπέρ κατά εγκρίνεται, συμβιβαστική AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική AM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 447 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 448 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 449 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική ZB υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική AM υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική EA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι η e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική e, F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 554 κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική CB υπέρ κατά υπέρ της συμβαστικής CB κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική CC με προφορική τροπολογία συμβιβαστική λοιπόν CC με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν χρειάζεται να φωνάζετε, μόνο να ψηφίζετε. Ε, συμβιβαστική λοιπόν χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική CD με προφορική τροπολογία πάλι από την ευθυντή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Χωρίς την προφορική τροπολογία η ίδια συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική CE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική CF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική CH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική CI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 594 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβαστική CJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική CL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική CM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 599 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική CP υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική TG υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 629. Πολλές σελίδες μετά. Μπερδεύτηκα λέει ο πρόεδρος. Πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβαστική AA Υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AB υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Συμβιβαστική SR ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική AD e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. S, συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Τροπολογία 720 υπερκατά κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική G Υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται. U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 71 έως 732 ομού υπέρ κατά αποχές απερίφθησαν. V συμβαστική υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται. W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική X υπέρ αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ή ε υπερκατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική αι υπερκατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική J υπερκατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική λ υπερκατά αποχές εγκρίνεται, Μ μη υπερκατά αποχές εγκρίνεται, n νη αποχές εγκρίνεται, 935 υπερκατά αποχές απερίφθη, συμβαστική Σ υπερκατά αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική Z, Z, α υπερκατά εγκρίνεται, α, ρο εγκρίνεται, 9, 27 υπερκατά απερίφθη, 988 υπερκατάποχε απερίφθη, 148 και ονομαστικά αρχιτεί ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 30 κατά. 25 υπέρ. Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, MA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AP υπέρ κατά αποχές. Α, DH. AP, λέει ο πρόεδρος. AP συμβαστική. Α, δεν το έχω αυτό. AP, έτσι, με προφορική, μάλιστα. Με προφορική, λοιπόν, δεν το είχα στο κατάλογό μου. Μα γιατί δεν το έχω εγώ. Οι ομάδες το έχουν υπόψη. Ο εισηγητής. or compromise AP? No, I have no oral amendment. No oral amendment. It was sent around. No. It came late. An oral amendment yeah, it came late, but I find very strange. Rapporteur is not a... Μπορεί να κατατέθει και μεγάλη καθυστέρηση, αλλά παράξενο μου φαίνεται να μην το ξέρει και ο εισηγητής, να μην το έχω και εγώ στον κατάλογό μου, τι συμβαίνει. So, you oppose, we oppose. So there is an opposition of the oral amendment. So we vote without the oral amendment. Uh, AP. Λοιπόν, ψηφίζουμε την AP σκέτη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική TH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία. 168. AG υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Y υπέρκατα αποχές εγκρίνεται. R ρο υπερκατά αποχές εγκρίνεται. C, Q υπέρκατα αποχές εγκρίνεται. 1088 υπέρ αποχές απερίφθη. Όμικρον υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 1092 και 93 Υπερκατά συγκρίνονται. εγκρίνονται 180 υπέρ αποχές απερίφθη 181 υπέρ απερίφθη F συμβαστική υπέρ εγκρίνεται P υπέρ εγκρίνεται 196 υπερκατά Ας το επαληθεύσουμε γιατί νομίζω ότι έχει απορριφθεί μένα αλλά ας γίνει έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. πέρας και απερίφθη. 197 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά απερίφθη. 198 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 199 και 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 281 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 285 ονομαστικά και αρχίζει Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 11 ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας. «206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 208 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 209 υπέρ, επαληθεύουμε, επαληθεύουμε την 209. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 210 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 14 υπέρ 14 κατά αποχές εγκρίνεται 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 227 υπέρ κατά επαληθεύουμε τη 227 227. Φαντάζομαι θα είστε αντίθετοι. Πέρας. Απερίφθη. Πρόταση της Επιτροπής αποστροποποιήθηκε ονομαστικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 45 υπέρ, 4 εις, ε, κατά 7 αποχές, εντολή για διοργανικές συνομιλίες, διαπραγματεύσεις, αρχής ψηφοφορία ονομαστικά, πέρας, 48 υπέρ, 7 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, στους σκιώδεις, τους συμβούλους και τη γραμματεία. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και συγχαίρω τους πάντες. Ήταν δύσκολο και περίπλοκο το θέμα. Έχουμε πλέον θέση της Επιτροπής λοιπόν και πλέον μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την αναγγελία στην Ολομέλεια ο τριμερής διάλογος, γύρι τριμερών διαλόγων, προφανές ε, σημάδι για τη βούλησή μας να ολοκληρώσουμε αυτό το πακέτο πριν από το τέλος του χρόνου. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή του Σκιώδης και όλους όσοι συνέβαλαν στο αποτέλεσμα αυτό. Και στο επόμενο θέμα μας έχουμε, αν μου δώσει κάποιος τον κατάλογο των ε, ε ψηφοφοριών, Ζήλε, ΒΑΤ, ε, ΦΠΑ, συγγνώμη, 41 όχι. Το Έλκιν υπέρ. Ωραία, υπερψηφίζεται λοιπόν. Επαληθεύουμε τη 41 ωστόσο. Τροπολογία 41 με επαλήθευση ηλεκτρονική. Πέρα στις φορείες. Παρακαλώ η ομάδα μου να μου δώσει τον κατάλογο των ψηφοφοριών για αυτή και την επόμενη ψηφοφορία. Ένα δεύτερο κατάλογο σας παρακαλώ. I I've been given only the banking. Okay, thank you. Uh, amendment 40... 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 43. Εναλλακτική συμβιβαστική α προφορική τροπολογία υπέρ κατά και επαληθεύουμε Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασα περίφθη. Ψηφίζουμε την αρχική εναλλακτική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά... Κατά ένα το μάλιστα. Ωραία. Επαληθεύουμε. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία 28-28, άρα περίφθη. Τα τρία υπέρ κατά απόχες. Επαληθεύουμε και πάλι. 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τ3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική β υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική γ υπέρ κατά ε, συμβαστική γάμμα, παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Α, είστε υπέρ. Όχι, τότε δεν χρειάζεται επαλήθευση. Εγκρίνεται λοιπόν. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60, 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εναλλακτική συμβαστική D δέλτα με προφορική τροπολογία υπέρ κατά και επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας και απερίφθη. Συμβαστική χωρίς προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ υπέρ υπέρ παρακαλώ κατά Απόχες απερίφθη. 69 υπέρ. Κατά. Απόχες απερίφθη. 16 υπέρ κατά αποχές. Όχι, να επαληθεύσουμε τη 16. Πέρας της ψηφοφορίας και έγκρινε η 17 τώρα παρακαλώ υπέρ κατά Καταλαβαίνω ότι δεν είσαστε σίγουροι, αλλά να επελθεύσουμε τώρα. Το 17 είναι μάλλον προς ισοψηφία Πέρας. Και εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. 28 υπέρ, 28, 27 κατά. 70 υπέρ κατά. Και επαληθεύουμε την 70. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία 28-28, άρα περίφθη. 18 υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε τη 18. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. Η 71 παρακαλώ υπέρ, κατά και επαληθεύουμε την 71. Πέρας. Απερίφθη. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 19 υπέρ. Κατά. Μάλλον ε, εγκρίθηκε, αλλά στο το επαληθεύσουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε, ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80-81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82-82 υπέρ κατά Μπορείτε παρακαλώ να κλείσετε το, την ψηφοφορία. Λοιπόν, επαληθεύουμε την 82 τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 82, καταπίπτει. 83 τώρα. Υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε την 83, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία άρα απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 84 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 85 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά επαληθεύουμε την 87 παρακαλώ αρχίζει ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική G υπέρ εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά απερίφθη, 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ. Για να επαληθεύσουμε την 27. Πέρας. Απερίφθη. 28 υπέρ κατά... Θα επαληθεύσουμε την 88, αλλά παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Πέρας και ισοψηφία. Απερίφθη δηλαδή. HE τα υπέρκατα αποχές εγκρίνεται, 32 υπέρκατα αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρκατα αποχές απερίφθη, 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 35 υπέρ αποχές απερίφθη, 36 υπέρ αποχές εγκρίνεται. Α, η γιώτα υπέρ αποχές εγκρίνεται, 39 υπέρ κατά και επαληθεύουμε την 39. Πέρασε ψηφοφορίας. Απερίφθη. Υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά. Και επαληθεύουμε την 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 40 σε τμήματα πρώτο υπέρ ΕΛΚ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρόταση στην πρόταση, ψηφοφορία στην πρόταση επιτροπής όπως τροποποιήθηκε ονομαστική παρακαλώ αρχής ψηφοφορία The vote is closed. 50... Πέρας της ψηφοφορίας 51 ψήφι 5, 2 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Ισηγητά. Περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση για το ε, επόμενο πρόγραμμα, τροπολογία 14. Θέλετε ε, κατάλογο ψηφοφορίας, ναι, θα περιμένω. So, amendment 14 in favor. μεταρρυθμίσεις ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός ε, A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά. Είστε κατά της προφορικής τροπολογίας της δικής σας. Εντάξει, απλώς ελέγχω. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την 44 με προφορική τροπολογία. Πέρα της ψηφοφορίας, 17 ψήφοι υπέρ, 35 κατά απορρίπτεται. Επομένως, αυτό ήταν η προφορική τροπολογία. Okay, we have to vote on four. Να ψηφίσουμε για το 44 χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση ξανά, άρχεται η ψηφοφορία. 44 χωρίς προφορική τροπολογία. Πέρας. Και απορρίπτεται ε, επομένως ε, υπέρ κατά αποχές ε, στις 45 απορρίπτεται, 46 απορρίπτεται, 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές ε, ε, απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 32 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση από της τροπολογίας 32 πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ονομαστική ψηφοφορία του τροποποιημένου κειμένου άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της, τροπο, της ε, ψηφοφορία 40 ψήφοι υπέρ 14 κατά μία αποχή. Και περνάμε επομένως στο, ε, στο σχέδιο προφορικής ερώτησης. Έτσι δεν είναι. Μαζί με ε, ψήφισμα για το IFF 17. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ψηφίσουμε on block, ομού, τις ερωτήσεις υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε ε, για το προσχέδιο ε, τροποποιημένης ερώτησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στο ίδιο το κείμενο του ψηφίσματος, τροπολογία 5, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν χρειάζεται νομίζω εδώ να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Άρα, τροπολογία 8, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αρχικό κείμενο παράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές κατά, κατά, νομίζω πως εγκρίνεται, λέει ο Πρόεδρος. Ηλεκτρονική επαλήθευση, πολύ ωραία, ε, για την 19, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας υπαριθμών 20 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 ψήφοι υπέρ, 25 κατά 2 αποχές. Ε, παράγραφος 9 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την τροπολογία 21, όχι ούτε... Ε, τροπολογία 22 λοιπόν απευθείας υπέρ κατά η ηλεκτρονική υπαλήθευση από της τροπολογίας 22 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές νομίζω ίδια πλειοψηφία. Εγκρίνεται. επομένω. τροπολογία 24 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 14 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 15 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο παράγραφος 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο παράγραφος 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 29 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο παράγραφος 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα από μου, ε, μαζί ε, μέχρι την 11 η τεολογική σκέψη τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο μου από την 13 μέχρι την 26 σκέψη υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Επίσης, ε, ABC αρχικό κείμενο τεολογικές σκέψεις κατά... Ε, αναφορές συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ε, ε, η F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Διολογικές αναφορές μέχρι την H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 4. Άρχεται. πέρας της ε, ψηφοφορίας ε, απερίφθη κείμενο, ψηφίζουμε τώρα με ονομαστική ψηφοφορία το τροποποιημένο κείμενο, άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας. 50 ψήφοι υπέρ, μία ε, ψήφος ε, εναντίον, τρεις αποχές, συγχαρητήρια. Και περνάμε Επομένως, μάλλον όχι, ολοκληρώσαμε, θα ε, σταματήσουμε για λίγο μια μικρή διακοπή περιμένοντας την κοινή συνεδρία των Επιτροπών ΕΚΟΝ και ΑΦΚΟ ε, που προβλέπεται στο σημείο 21. Λίγα λεπτά λοιπόν διακοπή παρακαλώ. Πέντε λεπτάκια. Γιατί αν έρθουν στην ώρα τους οι συνάδελφοι της ΑΦΚΟ θα περάσουμε μέσω στην ψηφοφορία. Στις 6.30 ακριβώς.